Welcome to the second part of this committee meeting. Uh, we'll now start with the first consideration of the draft. Λοιπόν, έχουμε την πρόταση γνωμοδότησης προς την πρωτοβουλία της ΕΤΡΑ, ΙΤΡΕ συγγνώμη, για την λεγόμενη κιανή οικονομία, έρευνα και ανάπτυξη στην κιανή οικονομία. Θα δώσω το λόγο στον, στην εισηγήτρια Λαουράγγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Αυτό το οποίο προσπάθησα να λάβω υπόψη στα πλαίσια της νομοδότησής μου είναι η σημασία της υπογράμμισης του ότι η οικιανή ανάπτυξη ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει την προστασία της θάλασσας. είναι απαραίτητο να διασωθούν και να, ανακτηθούν οι απώλειες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στους φυσικούς πόρους στα πλαίσια του πνεύματος της αηφορίας. Η αηφορία θα πρέπει να είναι κάτι το αποδεδειγμένο και βέβαιο. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί υφίστανται ανθρώπινες πιέσεις ιδιαιτέρως ισχυρές και δυσδιαχείριστες πλέον. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τεράστια προβλήματα για τις θάλασσες. Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα με τη μόλυνση, τις κλιματολογικές αλλαγές, τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν <clears throat> τις περιβαλλοντικές πλευρές του θαλασσίου περιβάλλοντος και να υπάρξει μια αρκιανή οικονομία, αηφόρος, βιώσιμη, η οποία όμως δεν θα περιορίζει και τις δυνατότητες απασχόλησης. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε λοιπόν αυτή τη λογική έτσι ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τους ωκεανούς και να βελτιώσουμε τις τεχνολογίες που έχουμε στην διάθεσή μας ιδιαίτερος όταν είναι έτοιμο να ενισχύσουμε, είμαστε, ε, είναι χρήσιμο να ενισχύσουμε την έρευνα η οποία θα έχει σαν στόχο ε, τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Για να ευνοήσουμε πράγματι την μπλε οικονομία, την κιανή οικονομία, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, είναι απαραίτητη η καινοτομία ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ναυπηγική βιομηχανία, οι υδατοκαλλιέργειες, οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η αλία. Και δεν θα πρέπει επίσης να αγνοούμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιβάλλον, το θαλάσσιο μέσα στο οποίο καλούμεθα να λειτουργήσουμε. Εγώ προσπάθησα να δω με ποιο τρόπο μπορούμε να <clears throat> βελτιώσουμε και τον λεγόμενο θαλάσσιο τουρισμό μαζί με τον παράκτιο τουρισμό. Είναι και αυτές οι μορφές τουρισμού σημαντικές για την ανάπτυξη την οικονομική και τη μείωση των προσωρινών ανασφαλών θέσεων απασχόλησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε πλήρη σεβασμό με το περιβάλλον. Η προστασία άλλωστε του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει ε, την δημιουργία θέσεων εργασίας και στα πλαίσια του περιβαλλοντικού τουρισμού. Ε, εγώ μιλάω για όριμο τουρισμό, για συνειδητοποιημένο τουρισμό, για πολιτισμικό τουρισμό ο οποίος να φέρνει στην επιφάνεια τον τομέα αυτό και κυρίως ένα σύγχρονο έτσι ώστε η δημιουργία θέσεων απασχόλησης να είναι κάτι το βέβαιο και υποστηρίξιμο χρονικά. Και τέλος προσπάθησα να αντιμετωπίσω και το θέμα της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου. Όλες οι πλευρές οι οποίες εμπλέκονται στην κοιανή οικονομία θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται στα πλαίσια ενός συνεχούς μονίμου και επικοδομητικού διαλόγου. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι όπως η κοινωνία των πολιτών, οι εργαζόμενοι κυρίως και οι επιχειρήσεις να συνεργαστούν, διότι μόνον έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό σωστά και θα το προστατεύσουμε σωστά. Και θα καταλήξουμε σε σημαντικές λύσεις οι οποίες θα έχουν κυρίως τοπική διάσταση σε μια πρώτη φάση. Λοιπόν, για να μέγιστοποιήσουμε την οικονομική αυτή και αηφόρο ανάπτυξη και για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ποιοτικού τύπου, είναι απαραίτητο να υπάρξει σωστή ανταλλαγή ε, των βέλτιστων λεγόμενων πρακτικών. Θα πρέπει η επιχείρηση, η έρευνα, η τεχνολογία να συνεργαστούν έτσι ώστε να προτείνουν λύσεις βιώσιμες και λύσεις ποιοτικές. Thank you. I'll give the floor. Θα δώσω το λόγο τώρα στους κοιόδης εισηγητές. Η κυρία Τζεντήλε πρώτη. Grazie, Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την εισαγωγή της κυρίας Τζέα συμφωνώ με την κατεύθυνσή της, ιδιαίτερα στον τομέα τον πολιτιστικό. Η θαλάσσια οικονομία αντιπροσωπεύει και θα αντιπροσωπεύει ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης και σωστής απασχόλησης. Χωρίς σε καμία περίπτωση όμως να μειώσουμε το ποιοτικό επίπεδο αυτής της πολιτιστικής αντίληψης. Η προώθηση της ιδέας της περιβαλλοντικής αηφορίας αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν πρέπει να απορρίψουμε. Μου φαίνεται επίσης σωστό να υπογραμμίσουμε το ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια σημαντική συνάντηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις από τη μία και την τεχνολογία και την έρευνα από την άλλη. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία των παράκτιων πληθυσμών και από την δυνατότητα την οποία έχουν δείξει να δημιουργήσουν νέα δίκτυα τουριστικά και πολιτισμικά συνδέοντας τις παράκτιες περιοχές και την θάλασσα με την ενδοχώρα. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης αγκυρωμένες στην παράδοση, οι οποίες όμως θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο από νέα περιεχόμενα και νέες αρμοδιότητες. Ε, Νομίζω ότι η Επίτροπη αυτή λοιπόν οφείλει να αποδεχθεί και ένα περαιτέρω ε, θα έλεγα χαρακτηριστικό των πολιτικών μας, τη θαλάσσια πολιτική, σαν ευκαιρία της κοινωνικής πολιτικής, σαν προώθηση της ισότητας των φύλων. Σαν ευκαιρία να προσφέρουμε στους πιο ευάλωτους ε, πληθυσμούς, όπως οι μετανάστες, όπως οι γυναίκες, όπως οι ανάπηροι, να μπορέσουμε να προτείνουμε σε όλες αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού την δυνατότητα κατάρτισης σε νέους τομείς και συνεπώς μια νέα ευκαιρία επανεισόδου στον κόσμο της εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ε, μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με ένα εγκάρσιο σχίσμα ανάμεσα στις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και στις δράσεις μας από την άλλη. Τώρα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να μην αγνοήσουμε έναν στόχο που θεωρώ σημαντικό, τον στόχο ο οποίος λέει ότι στο εσωτερικό της ε, βιοαϊφορίας περιλαμβάνονται και γεννιόνται νέες ευκαιρίες έτσι ώστε η Μεσόγειος να βγει από τη σκιά. Η Μεσόγειος να γίνει το κέντρο του προγραμματισμού μια σωστής επενδυτικής πολιτικής που θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η Μεσόγειος λοιπόν δεν θα είναι πια νεκροταφείο μεταναστών όπως δυστυχώς είναι και ήτανε και αυτές τις τελευταίες ώρες το είδαμε πάλι, αλλά θα είναι μια νέα ευκαιρία, όχι μόνο για την προώθηση πολιτικών ειρήνης, πολιτικών υποδοχής, αλλά και πολιτικών αποκατάστασης της αποστολής της Μεσογείου μέσα από την αλληλεία, μέσα από τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσα από τον τουρισμό και μέσα από την αποκατάσταση της ισορροπίας Βορρά και Νότου. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Τζεντήλε. Η Ούλα Τόρνες και σας ευχαριστώ που διευθύνατε τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Και τώρα είστε η σκιώδη συγγήτρια για την παρούσα έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε στα αγγλικά. Θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι η συγγήτρια συνέταξε ένα πραγματικά χρήσιμο σχέδιο για την γνωμοδότηση. Με ικανοποιεί η στόχευσή της στη βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην γαλάζια οικονομία, γιατί οι δεξιότητες αυτές επιτρέπουν και η πρόσβαση σε αυτές αποτελεί προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας. Και συμφωνώ με τη στόχευση επίσης της ε, συγκίτρια για την καλύτερη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων καθώς και ε, τρόπους μεταφοράς που να είναι πιο φιλικοί στο περιβάλλον. Ευχαριστώ την εισηγήτρια επίσης που τονίζει και τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στα πλαίσια της γαλάζιας οικονομίας που και αυτός μου φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Βέβαια μου λείπουν κάποια πράγματα στη γνωμοδότηση, βρίσκω να λείπουν και πρώτο μου φαίνεται σημαντικό να τονίσουμε τον ρόλο της ναυτιλίας όταν μιλούμε για γαλάζια οικονομία ιδίως την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τον τομέα της ναυτιλίας, καθώς βέβαια και το πώς θα πάει σχετικά με, την, με το σεβασμό του περιβάλλοντος ο τομέας αυτός. Επίσης, ο κλάδος δηλαδή, της ναυτιλίας. Να δούμε και τη μεγάλη δυναμικότητα που έχουν ε, οι πηγές ε, ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ νομίζω υπάρχει σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης και για μια πιο πράσινη Ευρώπη και η χώρα μου, η Δανία, έχει συλλέξει σημαντική εμπειρία στο τομέα αυτό. Θα υποβάλω τροπολογίες που θα τονίζουν αυτό το δυναμικό. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και πάλι την εισηγήτρια και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας πάνω στο κείμενο της γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ ο οποίος εκπροσωπεί πάλι με τη σειρά του τον σκιώδη συγητή του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αγέρα για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που αποτελεί ένα χρήσιμο έγγραφο που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Για την απασχόληση η γαλάζια οικονομία έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζόμενων που έχουν άμεση σχέση με την θάλασσα αλλά και με τις επιπτώσεις που έχει η γαλάζια οικονομία και στην ξηρά. Όσο αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γαλάζια οικονομία έχει το, τη δυνατότητα να δημιουργήσει 5,4 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης και σημαντικό τζίρο κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και να την καταστήσει αηφόρο, ιδίως με προώθηση του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις ιδιαιτερότητες του κάθε επίπεδου. Όπως είπε η κυρία Αγκοέρα, η συγκέντρωση στους φυσικούς πόρους και η καλύτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές είναι απαραίτητα για να γίνει βιώσιμη η γαλάζια οικονομία και για να προωθηθεί η δημιουργία απασχόληση. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πτυχές όπου θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Δηλαδή είναι ανάγκη να βελτιωθεί η γνώση για την κατάσταση του βυθού. Επίσης η γνώση αυτή να διαδοθεί καλύτερα να είναι καλύτερο συντονισμό του έργου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπή χωρών μελών και επιχειρήσεων του κλάδου με καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για να βελτιωθεί η κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα. Πρέπει να κατανοηθεί και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φυσικοί πόροι, να είναι γερά θεμελιωμένες επιστημονικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο της Ένωσης Χρειάζεται πιο ρεαλιστική γνώση, η οποία θα βοηθήσει να προωθεί και ανάπτυξη και η απασχόληση και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι αρμοδιότητες βέβαια είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Η γαλάζια οικονομία προσφέρει πολλές δυνατότητες και στην αλληλεία και στην ε, υδατοκαλλιέργεια, στη βιοτεχνολογία, στις επιστήμες των ωκεανών, καθώς και και μάλλον θα χρειαστεί όλα αυτά, θα χρειαστούν σε όλα αυτά άνθρωποι με ιδιαίτερε ε, γνώσεις και ικανότητες. Πρέπει να προωθηθεί ο τομέα αυτό και να ενισχυθεί η ελκυστικότητά του, ώστε και οι νέοι να προσελκυστούν προς τον ε, τομέα αυτό, προ τον κλάδο αυτό. Ε, θέλω να μιλήσω τέλος και για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό και όπως τα είπε και η συγχύτρια, είναι πολύ σημαντικός τουρισμός αυτός για πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και πρέπει να ενισχυθούν οι ε, θαλάσσιες δραστηριότητες. Έτσι θα επιτρέψουμε σε πολλές, ιδίω μικρέ και μέσες επιχειρήσεις και να αναπτυχθούν αλλά και να δημιουργήσουν απασχόληση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι Παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει το λόγο. Α, ο κ. Φρίσκ που είπατε δεν ε, ε, είναι παρόν. Είμαι ο Μάρκο Βάιντερ από την Γενική Διεύθυνση ε, Πόρων κλπ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγητία καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές για τις ενδιαφέρουσες ιδέες και την πολλή δουλειά που έχουν κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Σημειώνω ιδίως το ενδιαφέρον που δείχνεται για την απόκτηση δεξιοτήτων, καθώς επίσης και το περιβάλλον, καθώς και για τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης. Αυτά σημειώνω κυρίως και σε ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, τότε θα δώσω το λόγο ξανά στην κυρία για να ολοκληρώσει. Έχει το λόγο κυρία μου. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας, είναι σημαντική. Με βοηθά να εμβαθύνω και να εντάξω κάποια από τα στοιχεία τους στη δική μου πρόταση, εφόσον έχουν υπάρξει κάποιες ελλείψεις. Όταν μιλάμε για την κιανή οικονομία, μιλάμε για τουριστικές δραστηριότητες, προεχόμεθα από 28 χώρες, πολλές από τις οποίες εμπλέκονται άμεσα σε τουριστικές δραστηριότητες, κάποιες άλλες όμως όχι. Το να ενιοποιήσουμε δηλαδή αυτή την διαφορετικότητα των απόψεων είναι κάτι το σημαντικό. Ευχαριστώ λοιπόν την συνάδελφο Τζεντήλε θα σκεφτούμε αυτά τα οποία μας είπε, θα λάβουμε υπόψη μας τα οράματα τα οποία εξέθεσε επίσης και η συνάδελφος Ούλα Τόρνες στα πλαίσια της προσπάθειας έβρεσης μιας νέας ανανεωμένης ενέργειας για την παρέμβασή μας εδώ. Υπάρχουν δυνατότητες για συνεργασίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα με το οποίο θα συμφωνήσει η μεγάλη πλειοψηφία. Η συνεισφορά μας νομίζω θα είναι καθοριστική. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία είναι 22 Απριλίου, 12η Μεσημβρινή και η υιοθέτηση την 28η Μαΐου. Περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την κυρία Άγκια σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Για μία ακόμη φορά θα λώσω το λόγο στην κυρία Άγκια. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Έχω μεγάλο σουξέ, λέει η κυρία Άγκια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν πολλά προσφέρει στην προσπάθεια την οποία έκανα. Στα πλαίσια των συναντήσεων τις οποίες είχα με τους περισσότερους από τους εισηγητές, principale eh, focus quello di eh, ancora una volta una visione. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ομοιογένεια τις τάσει του Κοινοβουλίου σχετικά ε, με, ε, τα, με ε, το τι επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση αυτής της πρότασης επιστρέφοντας στο προηγούμενο έγγραφο του 2010. Το έγγραφο αυτό είδα πως ήταν διαρθρωμένο και συνειδητοποίησα ότι οι επιπτώσεις τις οποίες είχε στην καθημερινότητα ήταν ελάχιστες. Βασίστηκα επίσης ότι εκεί που το 2010 ε, θέταμε συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη, στη συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχουν αυτοί οι στόχοι. Και αυτό για μένα είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Προσπάθησα εγώ να επανεντάξω αυτά τα ε, στοιχεία Κάποιοι είπαν ότι η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι προηγήθηκε μια λαϊκή διαβούλευση. Οι πολίτες ε, έθεσαν τις ε, κατευθύνσεις οι οποίες απετέλεσαν τους στόχους της στρατηγικής αυτής. Πολλοί από τους στόχους αυτούς δεν έχουν γίνει ακόμα πραγματικότητα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανταλλάξουμε όλα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα και να τα κάνουμε καλύτερα. Προσπάθησα λοιπόν να αναλύσω λίγο περισσότερο την κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα της ανεργίας δυστυχώς, την οποία, η οποία μάλλον μαστίζει την Ευρώπη σήμερα βλέπουμε ότι προβλέπεται η έλλειψη απασχόλησης, η ανεργία σε διαφορετικά επίπεδα. Προβλέπεται επίσης και ο κίνδυνος της ένδυας σε ορισμένες χώρες. Υπάρχουν ορισμένες χώρες στις οποίες τα προβλήματα είναι οξυμένα Υπάρχουν χώρες στις οποίες όχι μόνο υπάρχει ο κίνδυνος της φτώχειας, αλλά υπάρχει η απόλυτη φτώχεια σε κάποια ποσοστά. Λοιπόν θα πρέπει να θεωρήσουμε την πρόταση αυτή όχι σαν μια διαπίστωση ήτας, αλλά σαν μια προσπάθεια για να κάνουμε ένα σημαντικό άλμα. Σημαντικό σημείο επίσης είναι η αναφορά η οποία γίνεται στα θέματα της φορολογίας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μεταφερθεί το βάρος από την εργασία σε άλλες μορφές στις οποίες το άχθος αυτό θα είναι, θα έλεγα, ελαφρύτερο. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να δούμε και ποιοι είναι οι φόροι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργούσαν λιγότερο τοξικά. Δεν θα πρέπει να είμαστε περιοριστικοί, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε στα κράτη τους τομείς τους οποίους μπορούν να βρουν καινοτόμες λύσεις έτσι ώστε να εξοικονομήσουν μεν χρήματα αλλά όχι στην απασχόληση. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις, την ισότητα των φύλων, την πράσινη απασχόληση. Φοβάμαι ότι δεν δίδεται σε όλα αυτά ιδιαίτερη σημασία τις κατευθυντήριες γραμμές του 2010 υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και σε συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ε, μιας και θα έλεγε κανείς ότι αφού δεν πετύχαμε ε, κάποια καλά αποτελέσματα σε ορισμένους τομείς, ε, τους βγάζουμε από τη μέση γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε αυτές τις κατηγορίες, τις κοινωνικές, που έχουν ανάγκη από καινοτόμες μορφές προστασίας. Αναγνωρίζουμε τις προτεραιότητες των κρατών μελών, αλλά δεν ξεχνάμε ότι εμείς εκπροσωπούμε την επιθυμία των πολιτών να προστατεύονται, να έχουν δομές υποστηρικτικές, οι οποίες να τους στηρίζουν εν πάση περιπτώσει. Το είπα λοιπόν νωρίτερα και το επαναλαμβάνω, ότι συνειδητοποιήσαμε ότι στα πλαίσια της ε, μετάφρασης των τροπολογιών μου σε άλλες γλώσσες, ε, δεν υπήρξε απόλυτα σωστή απόδοση της ιδέας την οποία εγώ θα ήθελα να προωθήσω. Η Γραμματεία έχει προωθήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις και εκεί όπου θα υπάρξουν οι διορθώσεις παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας το τελικό κείμενο έτσι ώστε να αξιολογήσετε σωστά λέγοντας ναι ή όχι στις προτάσεις τις οποίες εγώ κάνω. Η τελευταία πρόταση δηλαδή από πλευρά μου είναι η σωστή. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα είναι να μην αγνοήσουμε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης περισσότερο από άλλες επιτροπές έχει μια αντίληψη η οποία σέβεται τους πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. δεν έχει σημασία το ποιος υποβάλλει το συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μην κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα ξεχαστούν αύριο. Θέλουμε οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο, να λάβει υπόψη το Συμβούλιο το όραμά μας, διότι εδώ έχουμε μια έλλειψη οράματος. Εμείς προερχόμαστε όλοι περίπου από το χώρο της εργασίας. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ. Σκιώδης, εισηγητής του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Πρώτα για το έργο της εισηγήτριας, καθώς και για την συνεργασία της ήδη με τους σκιώδης εισηγητές δεν ε, μου φαίνεται άσχημη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού άπτεται όλων των σημαντικών θεμάτων όπως ε, κινητικότητα, εκπαίδευση, ελάχιστη μισθή, ε, η διτή μάθηση, η καταπολέμηση της και άλλα σχετικά θέματα. Χαίρομαι επίσης για την προσέγγιση που εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μετακινηθεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλους τομείς. Θα δούμε πού θα πρέπει να μετακινηθεί το φορολογικό βάρος. Υπάρχουν εκεί διάφορες σκέψεις, όπως για παράδειγμα περισσότερη επιβάρυνση της κατανάλωσης του κεφαλαίου ή της ε, επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Παρόλη την αισιοδοξία θεωρώ ωστόσο ότι ως κοινοβούλιο πρέπει να εγκύψουμε περισσότερο σε ορισμένα θέματα όπως τη μακροχρόνια ανεργία που είναι σημαντικό θέμα. Τους τελευταίους μήνες και χρόνια έχουμε μιλήσει πολύ για την ανεργία ιδίως των νέων που εξακολουθεί να παραμένει ένα καυτό θέμα. Χωρίς όμως να επιτρέπεται να λησμονούμε και τους μακροχρόνια άνεργους. Η μείωση της γραφειοκρατίας επίσης μου φαίνεται πολύ σημαντική, ιδίως για να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Η προώθηση τη κινητικότητα είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα και εδώ είναι σημαντικό να ε, ενισχυθεί το δίκτυο των διατάξεων της ε, απόσπασης εργαζομένων, να βελτιώσουν τη συνεργασία τους οι χώρες μέλη, να προσαρμόσουν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς τα εκπαιδευτικά του συστήματα και βεβαίως και τα συστήματα υγείας τους να λάβουν υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ψηφιακές κλπ. Οι στόχοι της στρατηγικής 2020 δεν επιτρέπεται να παραμεληθούν, όπως είπε και η συγκεκριά. Είμαστε ακόμα μακριά από οποιαδήποτε επίτευξη των στόχων αυτών και ιδίως ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας. Έτσι λοιπόν δεν επιτρέπεται να παραβλέψουμε την στρατηγική αυτή και τους στόχους της. Το ίδιο πρέπει να λάβουμε υπόψη επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες της νέας πολιτικής Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και που υποτίθεται θα οδηγήσουν στην επίτευξη στόχων του 2020. Είναι σημαντικό επίσης και συνεργαζόμαστε βέβαια επικοδομητικά στον φάκελο αυτό, γιατί μου φαίνεται σημαντικό να διατηρηθεί και η ταχύτητα με την οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις, ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις και να τις διαβιβάσει σύντομα στο Συμβούλιο, διότι αλλιώς φοβούμε ότι το Συμβούλιο δεν θα λάβει υπόψη του τις αποφάσεις μας, εάν δηλαδή για παράδειγμα δεν αντιδράσουμε αρκετά, αρκετά έγκαιρα. Ε, πιστεύω και νομίζω ότι και η η εισηγήτρια είναι σύμφωνη ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ δεν είναι πραγματικότητα ένα ευχολόγιο, αλλά συγκεκριμένε ξεκάθαρε προτάσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροδρίγε από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εργασία που επιτέλεσε η συγγετρία για πολλά θέματα για τα οποία θα πρέπει να καθορίσουμε τις καθεντήριες γραμμές με τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Για να αναφέρω κάποια, μακροχρόνια ανεργία, γι' αυτό υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ώστε να γίνει επανεκπαίδευση κάποιων ατόμων στην αγορά εργασίας για να βρουν μια νέα θέση απασχόλησης και μας ε, αρέσει και αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ για την ένδια και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε στα πλαίσια του δυνατού το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η ομάδα μας επιπροσθέτως θα καταθέσει τροπολογίες βελτιώσεων. Πρώτα απ' όλα για να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των κατευθυντηρίων γραμμών και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πράγμα το οποίο ανέλησε και η συγγήτρια και ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν, συμφωνούμε, και αποτελούν ένα εργαλείο, ένα μέσο της συνθήκης για να βελτιωθεί η στρατηγική μας του 2020. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του να αναφερθούν ρητός σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οι στόχοι της Ευρώπης 2020. Η απασχόληση, το ποσοστό φτώχειας και η εκπαίδευση οι στόχοι γύρω από αυτά τα θέματα. Επιπροσθέτως, προσθέτως, θα θέλαμε να προτείνουμε να τεθεί και ένας ειδικό στόχος για την ενεργεία των νέων εξαιτίας της ε, σημασίας που έχει το θέμα αυτό για την Ευρώπη. Δεύτερη βελτίωση που έχουμε κατά νου. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις διάφορες πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι για επιδείνωση των εργασι... συνθηκών εργασία τους και κοινωνικά ε, επιδεινώσεις αν θέλετε. Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρχει στις κατευθυντήριες γραμμές κάτι που να αναφέρεται στις πιέσεις αυτές οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Τρίτη βελτίωση, οι συντάξεις. Διότι για μας είναι απολύτως σαφές ότι αν θέλουμε Εμεί να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόληση. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, επαναλαμβάνω. Και όντω θα πρέπει να δούμε τι διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ της συντάξης και το σημερινό προσδόκιμο ζωή, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε διάφορες βελτιώσεις, γιατί αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας τελικά είναι ε, τα χρόνια κατά τα οποία συνεισφέρει στα κοινωνικά συστήματα ο κάθε εργαζόμενος. Πρόκειται για ένα πρωταρχική σημασία θέμα για να δούμε πώς θα εξασφαλιστεί το ότι τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια και εξήγηση επί αυτού του θέματος κατευθυντήρης Σε Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κύριος Κλασαντεύσκη, TCR. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας δίδει την δυνατότητα να κάνουμε σε αυτό το πρώιμο στάδιο ανταλλαγή απόψεων. Είναι ενδιαφέρον για μας, παρά το γεγονός ότι είμαστε από διαφορετικές χώρες και έχουμε διαφορετικές πολιτικές, ότι οι απόψει μας συμπίπτουν για τα οικονομικά και τα κοινωνικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη και την κατάσταση σε αυτούς τους δομείς που επικρατεί στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι παρήλθε η εποχή την οποία η οικονομική πολιτική εξεταζόταν μόνο από την άποψη την χρηματοπιστωτική. Το κοινωνικό ε, πρόβλημα είναι μεγάλο. Στα πλαίσια της ε, οικονομικής πολιτικής λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν ε, ε, σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό το κοινωνικό σκέλος της οικονομικής μας πολιτικής. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κοινέ θέσεις και αυτό το οποίο μου αρέσει είναι το ότι η συγγήτρια υπογράμμισε την ανάγκη να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάτι το οποίο επίσης ελέγχθη που είναι το θέμα της φορολογίας σε πολλές χώρες, της φορολόγησης της εργασίας σε πολλές χώρες που είναι επαχθής. Θα πρέπει η αγορά εργασίας να είναι συμπεριληπτική. Ειδικέ προτάσεις λοιπόν τις οποίες κάνετε για το θέμα αυτό και οι λύσεις που προτείνετε πιστεύω ότι είναι πολύ καλές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει και για αυτό το δικό σας έγγραφο και άλλα έγγραφα στα οποία αναφερθήκατε και πιστεύω ότι παντού θα πρέπει να μιλούμε για την οικονομική ποικιλομορφία της Ευρώπης, γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική από μία χώρα της Ευρώπης και σε άλλη και οφείλεται και εν μέρει στο γεγονός ότι οι οικονομίες των κρατών μελών έχουν διαφορές αλλά έχουν και κοινά σημεία. Άρα θα πρέπει όλες οι προσπάθειες και δραστηριότητες να συντονίζονται στα πλαίσια αυτών των διαφορών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά ε, νομοθετικά πλαίσια, διαφορετικές συνθήκες ζωής, αλλά θα τα πρέπει να τα θυμόμαστε αλλά και να συντονίζουμε τις προσπάθειές μας. Το κοινωνικό dumping εκείνη επίσης αναφέρεται. Άρα γενικά έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε ακόμη και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε για τα σημαντικότατα αυτά θέματα σε συμβιβαστικέ λύσεις και προτάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Βέμπερ. Από Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις απόψεις που εκφράζει για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε αυτό το σημαντικό θέμα, το ότι ε, ήρθε σε επαφή με τις ε, σκιώδεις εισηγητές ε, και σέβεται τις απόψεις των άλλων και θα αντικατοπτρίσει τις απόψεις όλων. Έχουμε συμβουλευτικό ρόλο το θέμα αυτό και βάσει προηγουμένων εμπειριών επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το πόσο μπορούμε αυτή τη στιγμή να επηρεάσουμε το Συμβούλιο στις αποφάσεις που λαμβάνει. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι σημαντικό μέσω αυτών των εκθέσεων και μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση να στείλουμε μήνυμα για να ξέρουν οι πάντες ποια είναι η άποψη αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ίσω κάποια στιγμή αργότερα θα ληφθούν υπόψη. Βεβαίω εξυπακούεται ότι Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών της απασχόλησης και της στρατηγικής του 2020. Γι' αυτό θέλουμε να ε, εστιαστούμε και στην αναθεώρηση αυτής της στρατηγικής. Συμφωνούμε με πολλές από τις απόψεις και την προσέγγιση που εξέφρασε η συγγήτρια και την υποστηρίζουμε βεβαίως Πρέπει να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις. Υποστηρίζουμε την ιδέα των οικογενειακών επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τους μακροχρόνια ανέργους. Θέλουμε συγχρόνως να τονίσουμε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Είναι σαφές από την έκθεση της Επιτροπής και επιμένουμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή όταν συζητώνται τέτοιου εκθέσεις να είναι παρούσα για να μας δίδει ακριβώς την σαφή εικόνα των αναγκών της αγοράς εργασίας και να μας δίνει την πλήρη εικόνα της οικονομίας, ότι χρειάζονται τέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης. Και βεβαίως η κατάρτιση, επανακατάρτιση και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά και οι λιγότερο εξειδικευμένες εργασίες είναι απαραίτητες στην Ευρώπη και υπάρχουν άτομα τα οποία θα κάνουν αυτές τις εργασίες. Ένα ιδιαίτερο θέμα για το οποίο θα, στο οποίο για το οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι ότι η κοινή αγορά της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι είναι πραγματικότητα όσον αφορά την ενδοκινοτική ε, κινητικότητα και σήμερα τα σύνορα ακόμη και στην αγορά απασχόληση δεν είναι τα ίδια όπως παλιά. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας και να προετοιμάσουμε αυτούς που αναζητούν εργασία να την αναζητήσουν και άλλες χώρες πλην της, εκτός της πατρίδας τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συστάσεις εκ μέρους Επιτροπής προς τα κάτι μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις γειτονικές χώρες του καθενός και τις χώρες τις οποίες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μετακίνηση εργαζομένων Προ άλλε Θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα οποία πραγματικά ζητά η οικονομία και η αγορά εργασία. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική αρρωγή, πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να καταλήξουν σε κατάσταση ένδυας εάν οι γονείς τους είναι μακροχρόνια ανεργία. Διότι αν δεν κάνουμε τις κατάλληλες επενδύσεις αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν αυτή την οικογενική τους παράδοση πλέον που θα έχει γίνει η ανεργία και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Αλλά βεβαίως όλοι υποστηρίζουν έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λάμπερτ. για τους πρασίνους έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ την σκιώδη μας, την κυρία Ζενόφκα εδώ. Θα ήθελα να πω πόσο θετική βρίσκουμε την έκθεση, η συγγήτριά μου. Ε, κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και σαφώς και εκτιμούμε ε, την υπογράμμιση του προβλήματος της φτώχειας και της ανάγκης αποκατάστασης των συμμετριών. Δεν υπάρχει συν απόφαση για τις κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχει δυστυχώς απλή διαβούλευση και για μια ακόμη φορά μας ζητείτε να το κάνουμε αυτό με πάρα πολύ υψηλή ταχύτητα. Αν και είχαμε την ελπίδα ότι για μια φορά τουλάχιστον θα είχαμε την δυνατότητα να μας διαβουλευτούν λίγο νωρίτερα και να μας δώσουν περισσότερο χρόνο. Πάντως γενικά είναι μια καλή έκθεση. Ε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι θα έλεγα αρκετά απροσδιόριστες και γι' αυτό και υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες Έχουμε κάποιες ανησυχίες και στο κράτος μέλος το οποίο εκπροσωπώ υπάρχουν αρκετές νέες θέσεις, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις ενώ πληρώνονται στη δουλειά τους γιατί δεν επαρκούν τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Προφανώς και κάτι πρέπει να γίνει εδώ, όπως επίσης και θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία των στοχευμένων επενδύσεων που δημιουργούν απασχόληση Αρκετά μέλη έθεσαν επίσης μέσω των τροπολογιών τους το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας. Προφανώς εμείς θα πρέπει να είμαστε υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης σαν κλειδί της στήριξης των μεταβατικών περιόδων από τις οποίες περνούν οι πολίτες εφόσον χάσουν την δουλειά τους και αναγκαστούν να εργάζονται σε προσωρινή βάση και θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και κάποια στοιχεία για την έλλειψη και καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Πολλοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους λόγω ακριβώς διακρίσεων τις οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει μία παρατήρηση, όχι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, ο κύριος Γιούφτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια και τις συνεισηγήτριες για την προσπάθεια την οποία έκαναν και θα λάβουμε υπόψη τις προτάσεις τους. Και επιστρέφω στην κυρία Άγκια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Τις προτάσεις τις είχα ακούσει και στις συναντήσεις τις οποίες είχα μαζί τους και στις μελλοντικές συναντήσεις θα τις ε, ε, ακούσω εκ νέου και θα τις λάβω απολύτως υπόψη. Θα προσπαθήσω να καταστήσω τους στόχους μας ε, κάτι το οποίο να συμμερίζονται όλοι, χωρίς διαφοροποίησεις. Σας ευχαριστώ που εμείνατε και στα θέματα, προβλήματα της ανεργίας της μακροπρόθεσμης. Το θέμα της ε, διαχείρισης του εξαμήνου είναι ένας από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση προθέσεων είναι κάτι το θετικό και μπορεί να επηρεάσει θετικά και τις δικές μας προτάσεις. Πολλά μένει να γίνουν στις επόμενες συναντήσεις με τους κοιόδης. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις διαφορές εκεί όπου υπάρχουν σε επίπεδο απόψεων και έτσι να ακουστεί η φωνή μας και όχι μόνο η δική μας φωνή αλλά και η φωνή όλων των πολιτών που μας έστειλαν εδώ. Σας ευχαριστώ κυρία Άγκια, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 22 Απριλίου απόγευμα, 26 Μαΐου εξέταση τροπολογιών και 16 Ιουνίου υιοθέτηση, ψηφοφορία δηλαδή. Περνάμε τώρα στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για το έγγραφο εργασίας σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργή γύρανση και την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενναίες. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουκάν. Ο κύριος Κουκάν δεν είναι εδώ. και δεν υπάρχει φαίνεται ότι κάποιος, ε, δεν υπάρχει μάλλον κάποιος που να αντικαθιστά τον κύριο Κουκάν και θα δώσω τώρα το λόγο στην σκιώδη εισηγήτρια των σοσιαλιστών την κυρία Μπίλη Τσινκιούτε kuris e, galėtų būti mūsų geras pagrindas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας έχουμε ήδη συζητήσει. Ευχαριστώ για τη συζήτηση μέχρι τώρα και έχω να τονίσω ορισμένα θέματα. Θεωρώ ότι στην έκθεσή μας πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για την αξιολόγηση αυτού του ευρωπαϊκού έτους, δηλαδή σχετικά με τα κριτήρια, πρέπει ιδίω να πούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική αυτή και να αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω. Και ποιες αποφάσεις οφείλουμε να λάβουμε για την πολιτική αυτή. Το έτος αλληλεγγύης προς τους ηλικιωμένους αξιολογήθηκε θετικά. Αυτό είναι καλό. Και ιδίω αξιολογήθηκε θετικά διότι απέδωσε και με μικρότερη χρηματοδότηση από ότι το προηγούμενο που ήταν το 2011. Το έτος αυτό μπορεί να γίνει εφαλτήριο για άλλες δραστηριότητες για την πρόθεση της αλληλεγγύης στον τομέα αυτό και ιδίω εν ώψη των δημογραφικών εξελίξεων και των μελλοντικών προοπτικών οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι είναι γεγονός η γύρανση της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι και τις μεγαλύτερη ηλικία να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αλληλεγγύης βάζοντας έτσι το θεμέλιο για το μέλλον. Αυτό καλούμεθα να κάνουμε. Τώρα έχω και ένα άλλο θέμα που είναι η ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην επαγγελματική ζωή. Πρέπει να συνεχιστεί η ενεργό συμμετοχή του στην επαγγελματική ζωή. Γιατί αντιμετωπίζουμε και ανεργία των ε, μεγαλύτερων ηλικιών. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους και πρέπει να μετεκπαιδευτούν. Πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο με τους εργοδότες, ώστε οι εργοδότες να λάβουν κίνητρα για να επενδύσουν στους ε, πλέον ηλικιωμένου και στο μέλλον τους. Στην έκθεση βέβαια περιλαμβάνεται και ότι οι στόχοι που είχαν βάλει το 2012 δεν επιτεύχθηκαν. Τονίζω ότι η διοργάνωση του έτους το 2012 περιλάβαν κυρίως συμμετοχή ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ούτως ή άλλως στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσπάθεια στο μέλλον με ειδικέ δράσεις να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε προστιθέμενη αξία και να διευρύνουμε τις δράσεις αυτές. Γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να, είναι, ε, να διευρυνθούν οι δραστηριότητε και πρέπει να μιλήσουμε και για την αηφορία όχι μόνο τους, των συνταξιοδοτικών συστημάτων αλλά και των συστημάτων υγείας. Ο εισηγητής τα λέει αυτά και στο εγγραφό του. Εγώ όμως έχω να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα γιατί βρισκόμαστε τώρα μετάσταση που το 2004 όταν εντάχθηκαν οι χώρες μας τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Λιθουανία, την χώρα μου, τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ένα πρόβλημα. Ότι δηλαδή πολλοί νέοι άνθρωποι καλά καταρτισμένοι σηκώθηκαν και έφυγαν από την πατρίδα μας και πήγαν σε άλλες χώρες μέλη. Στο μέλλον αυτό θα οδηγήσει όμως σε σημαντική πίεση στα κοινωνικά μας συστήματα, διότι θα λείπουν οι άνθρωποι αυτοί. Αφού οι πιο ενεργοί και καλά καταρτισμένοι άνθρωποι σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Έχουμε όμως την εφεδρεία των πλέον ηλικιωμένων που μπορούν να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η φορεία των συστημάτων. Πρέπει βέβαια να επενδύσουμε σε ζητήματα όπως η πρόληψη των ασθενειών, η καλή υγεία, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Και όλα αυτά να γίνουν πιο προσβάσιμα, πιο προσιτά. Ώστε και στην καθημερινή μας ζωή να μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο για τις στις υποδομές εκείνες που είναι χρήσιμες και απαραίτητες για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή, θα υποβάλουμε και κατάλληλες προτάσεις και τροπολογίες και σε ευχαριστώ εν τέλει πολύ. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Α, ο κύριος Κούκαν. Πέστε μας παρακαλώ, ο συζητητής, ακούσαμε την πρώτη σκιώδη εισηγήτρια διότι βέβαια έχουμε προχωρήσει κάπως ταχύτερα. Όμως τώρα σας δίνω το λόγο. Ε, έχει έρθει η σειρά σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. μεγάλη ευχαρίστηση σας παρουσιάζω το έγγραφο εργασίας για την 2012 ε, το Ευρωπαϊκό του Ενεργού Γέρνησης και Αλληλεγγύη μεταξύ γενναίων. Πρόκειται για την πρόκειται έκθεση που παρουσιάζω στην Επιτροπή Απασχόλησης. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία για μένα το θέμα αυτό, διότι κοιτάζοντάς με θα δείτε ότι εγώ είμαι ένα ενεργός γυράσκων και θέλω να παραμείνω ενεργός και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το μέλλον της Επιτροπής. Τι πραγματεύεται κυρίως η εκθεσή μου. Θέλουμε να αξιολογήσουμε το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε εκείνη το 2012 και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία όχι μόνο για να δούμε τι έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα, αλλά να συνεχίσουμε και την συζήτηση προσβλέποντας το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω και συστάσεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Για να απλούστο το λόγο. Εμείς στην Ευρώπη ζούμε περισσότερο, έχουμε λιγότερα παιδιά και η γυριά μας Ήπειρος αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλη δημογραφική αλλαγή. Οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται, η οικονομία αλλάζει και το πρόβλημα των γενεών υπάρχει. Θα αρχίσουν τα πράγματα λοιπόν να είναι πιο ε, σημαντικά από το 2000 2015-2035 ε, όταν οι baby boomers και όσοι γεννήθηκαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται και να αποσύρονται. Και το 2010 Μάλλον θα απλοποιήσω. Υπάρχουν τέσσερι εργαζόμενοι, υπήρχαν τέσσερι εργαζόμενοι για ένα συνταξιοδοτούμενο. Το 2020 θα έχουμε δύο εργαζόμενους για έναν συνταξιοδοτούμενο. Η κατάσταση λοιπόν θα αλλάξει άρδιν. Η ενεργός γύρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών είναι ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει όλοι από κοινού να βρούμε λύση. Δεδομένου ότι εδώ υπάρχουν και διάφορα θέματα κοινωνικής πολιτικής ε, οικονομικής πολιτικής, πολιτικής απασχόλησης, δημόσιας υγείας κτλ. Όχι μόνο γυράσκει η Ευρωπαϊκή πυρός, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών και διαφόρων περιοχών. Και πολλές φορές οι διαφορές αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες το 2012 με το ευρωπαϊκό αυτό έτος έγινε προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι πάντες τι σημαίνει ενεργός γύρενση και να γίνουν συζητήσεις ώστε να μπορέσουμε να ξεύρουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να προωθήσουμε δραστηριότητες κατά των στερεοτύπων, της, των διακρίσεων υπέρ των μεγάλων ανθρώπων σε ηλικία και θα ήθελα να αναφέρω ότι το θέμα αυτό συμπεριλήφθη στην μερίσια διάταξη των συζητήσεων που γίνονται σε κάθε κράτο μέλος. Πρώτα απ' όλα για να μπορέσει η συνειδητοποίηση των πάντων να, για το θέμα αυτό να γίνει σε όλα τα επίπεδα εθνικό και ευρωπαϊκό. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες ενεργού ε, γύρενσης και διάφορες πράγματα που λέγονται για την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων γενεών. Αυτό το θέμα απασχόλησε πολύ τα μέσα ενημέρωση, το σχολείο κτλ. Παρά το γεγονός ότι ο διάλογος στην πολιτική αυτή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γύρες του 2012 ήταν επιτυχής, δεν έγινε δημιουργήθηκαν νέα δίκτυα συζητήσεων, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων δεν ήταν ομοιόμορφη και οι επιχειρηματίες δεν ε, ενδιαφέρθηκαν από το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει επανεξέταση των πολιτικών των σχετικών σε κάθε επίπεδο και οι βέλτιστες πρακτικές να μπορέσουν να, να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Όλα αυτά ώστε να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα αυτό που θα κάνουμε. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες, να ενισχυθεί η, η γνώση και η εξειδίκευση αυτών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά των διαφορών γενναιών βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του έτους αυτού 2012 ε, επεκτείνονται και πέραν των ετών αυτών και κάποια θα είναι βιώσιμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνάδελφοι, θα πρέπει τον γυράσκοντα πληθυσμό μας να τον δούμε ως ευκαιρία αντί για βάρος οι συστάσεις μου θα εστιάζονται σε συγκεκριμένα θέματα και θα αφορούν κυρίως τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει διάφορα επιτυχή προγράμματα να εφαρμοστούν και να γίνει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Και επί αυτού του θέματος έχουν ε, τεθεί σε κίνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάφορες πρωτοβουλίες στα πλαίσια αυτού του έτους θα πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει οι επαφές μεταξύ των διαφόρων σχετικών δικτύων να συνεχιστούν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο συντονισμός μεταξύ αυτών που κάνουν τις διάφορες πολιτικές σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών και αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις να είναι πιο εντατικές. Θα πρέπει οι πολιτικοί, οι, εκπρόσωποι των ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι της τρίτης ηλικία, οι επαγγελματίες τεχνολόγοι από κοινού να συζητήσουν κάποια πράγματα. Το να αναπτύξουμε την αργυρά οικονομία είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να λαμβάνουν υπόψη οι ανάγκες του γυράσκοντος πληθυσμού και να ληφθούν υπόψη τα ειδικά, ειδικές ανάγκες, οι ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας και να ληφθούν όλα αυτά τα θέματα υπόψη από τον εμπορικό τομέα, από τον οικονομικό τομέα και υπόψη στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Η ενεργός ε, ε, γύρανση είναι μια πραγματικά για όλους και η κοινωνία θα πρέπει να λάβει με υπόψη το γεγονό ότι αυτά τα άτομα είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας και θα πρέπει να υποστηριχθούν στην καθημερινή του ζωή. Οι νέες γενιές θα πρέπει να αν διαφορθούν το θέμα αυτό και ο διάλογος μεταξύ όλων των γενναιών να ενθαρρυνθεί. Επίσης, να υπάρξει ειδική εστίαση στο γεγονός της διαβίου μάθησης δεδομένου ότι δίδενται έτσι περισσότερες ευκαιρίες στο του πληθυσμό να έχει καλύτερες δυνατότητες απασχόλησης. Τέταρτον, να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και τις διακρίσεις τις ε, ηλικιακές. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχείς πολιτικές στον τομέα αυτό, θα πρέπει να μην έχουμε πλέον διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία. Και εγώ δεν σας ομιλώ όσον αφορά μόνο την πρόσβαση σε θέση εργασίας στην αγορά εργασίας, αλλά και στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των ατόμων, όλων των μελών αυτής της κοινωνίας μας, που κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν ευάλωτα, να γίνουν αντικείμενο καταχρήσης και θα πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερως. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μία παράθεση από το Ευρωπαϊκό Αυτό έτος 2012. Η ενεργός γύρενση σημαίνει ότι γερνάει κανείς με καλή υγεία ως πλήρες μέλος της κοινωνίας του, αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση στη δουλειά του, πιο ανεξάρτητος στην καθημερινή του ζωή και συμμετέχει περισσότερο στα στα θέματα της πολιτείας. Προσπαθώ στην έκθεσή μου να αντικατοπτρίζονται όλες αυτές οι ιδέες και να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να συνεχίσουμε στα πλαίσια του έτους που αναπτύχθηκε το 2012. Συνάδελφοι, προσβλέπω στην συνεισφορά σας. Συζητούμε τώρα για πρώτη φορά το έγγραφο εργασίας και θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους της ε, ε, διαπολιτικής ομάδας για την ενεργό γύρεση επίση να μου αποστείλει σχόλια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you and you are really... Ευχαριστώ πολύ. Λέτε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ενεργοί ακόμα και σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία και άκουσα σήμερα για μια γυναίκα 67 ετών φανταστείτε που θέλει να γίνει πρόεδρος των Ενωμένων Πολιτειών. Αλλιώ ήταν τα πράγματα πριν από 50 ή 75 χρόνια, έτσι δεν είναι. Κρασνοντεύσκη τώρα είναι ο επόμενος και ο που λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα αυτά βέβαια είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε στην πολιτική μας ομάδα μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με δημογραφικά θέματα, με τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και τη γύρανση της κοινωνίας ε, της Ευρώπης. Όταν δεν ήμουν ακόμη Ευρωβουλευτής ήμουν απλά ενεργός πολίτης στη χώρα μου, χώρα μέλος της Ένωσης, δεν διεπίστωσα και μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο έτος 2012 και στα άλλα έτη, σε ό,τι αφορά δηλαδή και την δραστηριότητα των πλέον ηλικιωμένων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών. Ίσως να υπήρξαν τέτοιες ε, εξελίξεις ίσως πράγματι να είχαν κάποια επίπτωση στις κοινωνικές πραγματικότητες αλλά αμφιβάλλω. Πάντως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε υψηλότερε ηλικίε συνταξιοδότηση. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το σωστό. Μιλήσατε για την υποψηφία για την Προεδρία στις ΗΠΑ, Πολιτείες, αλλά υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα ανθρώπων που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ε, σε μεγαλύτερη και άκουσα για τη Γερμανία, στην Γερμανία μάλλον, για μια 65 άρισα η οποία περιμένει πεντάτημα. Ε, κοιτάξτε, βέβαια πρέπει να αλλάξει η στάση απέναντι στους ε, ηλικιωμένους. Εάν κάνουμε τη σύγκριση με τις ΗΠΑ και με, μεταξύ αυτών δηλαδή και των χωρών μελών της Ένωσης, Η γύρανση είναι εντονότερη στην Ευρώπη. Να σας πω τώρα για κάτι το οποίο δεν έχει περιληφθεί μέσα στο σχέδιο εκθέσεως και το πρώτο βέβαια ήδη αναφέρθηκε στην συζήτηση. Η δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων δεν μπορεί να αποτελεί υποχρέωση, ούτε μπορεί να τους επιβληθεί έτσι ώστε να λυθούν κάποια οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο αυτό συμβαίνει συχνά. Συχνά η βιολογική ηλικία των ανθρώπων σε διάφορες χώρες εξαρτάται και από τις κοινωνικές συνθήκες που ισχύουν στις χώρες αυτές ε, έχει πολύ, διαφορετικές, πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Σε ορισμένες χώρες οι ηλικιωμένοι έχουν καλύτερη ή χειρότερη πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, η αξιοπρέπεια του ηλικιωμένου και πολύ συχνά και η κοινωνική συμπερίληψη προκύπτει και μέσα από την συμμετοχή τους στην οικογενειακή ζωή. Το να καταστούν πιο ενεργά τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποξένωσή τους από την κοινωνία. Αυτά ωστόσο είναι καμιά φορά συνέπειες των εξελίξεων της αγοράς κλπ. Έχω και ένα γλωσσικό σχόλιο. Αυτό το active aging όπως το λαμβάνουμε από τα αγγλικά. Πάντως αυτό, αυτή η ενεργός γύρανση στα πολωνικά τουλάχιστον μου φαίνεται ένα γλωσσικό τέρας. Ε, σημαίνει ίσως να δραστηριοποιήσετε σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά στα πολωνικά δεν, δεν ηχεί καθόλου καλά. Ίσως θα πρέπει ε, να, πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε τη διαδικασία γύριανσης. Τι να πω, να γίνουμε νεότεροι. Ε, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει να φτιάχνει περίεργες φράσεις, αλλά Ελπίζω τέλο πάντων αυτό, αυτή η ενεργό γύρανση, ε, όπω διατυπώνεται στα πολωνικά, να βρει κάποια καλύτερη μετάφραση. Βάγκελ, ε, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος συνάδελφος στον οποίο να ήθελα να ε, αναθέσω την σύνταξη της έκθεσης αυτής από τον συνάδελφό μας που την έχει αναλάβει. Να έρθω σε αυτό που είπε ο Πολωνός συνάδελφός μας προηγουμένως. Και εγώ διαφωνώ με την ιδέα της ενεργού γύρανσης. Προτιμώ την παθητική γύρανση, έτσι ώστε να κρατήσει και περισσότερο. Ε, τέλος πάντων κάποια στιγμή όλοι θα φτάσουμε βέβαια στην ηλικία αυτή. Πάντω κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Αυτό είναι γεγονό. Νομίζω επίσης και μπορώ να πω ότι είμαι και βέβαιος ότι η έκθεση που θα συνταχθεί εν τέλει θα είναι πραγματικά καλή. Όταν ο νεοεκλεγή πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε το πρόγραμμά του, εγώ ρώτησα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές αλλαγές. Ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση. Ελπίζω ωστόσο ότι έχει σημειώσει την ερώτησή μου και ότι και ότι τα μέλη της, ε, των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών είναι διατεθειμένα να συζητήσουν το θέμα και να το προωθήσουν στο μέλλον. Βλέπω, ότι, βλέπω σήμερα μάλλον ότι συχνότερα από ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία που ε, συμμετείχα συζητούμε την ενεργογύρανση. Αυτό γίνεται και υπό το φως των διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών πτυχών. για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γέρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ γενεών, εγώ σημειώνω την πληροφορία ότι μόνο 42% των Ευρωπαίων πολιτών ενδιαφέρονται για την μοίρα των ηλικιωμένων. Παρόλο που πολλοί από αυτούς ήδη συναποτελούν μέρος αυτής της γενιάς αλλά πιστεύω ότι πολλοί δεν βλέπουν τους εαυτούς τους ως ανθρώπους που ε, γυράσκουν. Γιατί βέβαια το ποσοστό θα έπρεπε να είναι περισσότερο από 42%. Πάντως, πιστεύω ότι με την συζήτηση της εκθέσεως και του θέματος θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να λάβει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης προς την κατεύθυνση της θέσπισης σύγχρονων μέτρων για την ενεργογύρανση. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε προγράμματα για την απασχόληση των νεότερων ηλικιωμένων οι οποίοι γίνονται καθίστανται άνεργοι μέσα σε περίοδους κρίσεων και έχουν ακόμα διάθεση να ε, εργαστούν. Πρέπει να προωθήσουμε σχετικά μέτρα. Είναι και μερικά πράγματα τώρα που έχουν σχέση με την προστασία της υγείας και όπου οι σχετικές προδιαγραφές και πρότυπα θα πρέπει να εναρμονιστούν με προσπάθεια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλο θέμα που με απασχολεί πολύ είναι εάν μπορούμε ίσως να θεσπίσουμε ενιαία πρότυπα και να θεσπίσουμε και μια εποπτεία επί των συνταξιδοτικών ταμείων. Πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα συνταξιδοτικά ταμεία για να καλύπτουν τα κενά που έχουν στους προϋπολογισμούς των χωρών τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Βρίσκω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό και ότι χρειάζεται να μας απασχολήσει περισσότερο. Τελειώνοντας να πω δύο λόγια για το πώς μπορεί ο πληθυσμός που γυράσκει να βοηθήσει άλλους. Στη Σλοβενία, τη χώρα μου, έχουμε σχετικά παραδείγματα. Έχουμε 600 εθελοντές περίπου, οι οποίοι φροντίζουν 150.000 ακούμε, άλλους επίσης ηλικιωμένους, εξασφαλίζοντας τους μια ποιότητα ζωής. Ίσως πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να αναγνωρίσουμε αυτή την υποστήριξη που προσφέρουν ηλικιωμένοι άνθρωποι σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Και να ενισχύσουμε και μια υποστήριξη επαμοιβή. Κάνοντας την έτσι και επάγγελμα ή έστω ε, μια ε, παράπλευρη δραστηριότητα εφόσον έχουν κάποια άλλη απασχόληση. Οι χρονιές που έχουν περάσει παλαιότερα και αποκρίθηκαν έτος τάδε, έτος δίνα και εκείνο το περίφημο έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ διαφόρων ομολογιών ή μεταξύ ε, διαφόρων θρησκευτικών μειονοτήτων δεν απέδωσαν μπίζωνα αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος τα πράγματα θα πάνε διαφορετικά και θα υπάρξουν πλέον αποτελέσματα διαρκή και θετικά για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ευχαριστώ. οι σκιώδεις για την ΚΟΕ και τους Πρασίνους και το FDD δεν είναι εδώ, οπότε όποιος έχει ζητήσει το λόγο... Η κυρία Γιαζοβλέσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Γνωρίζω πάρα, πολύ, πάρα πολλούς οι οποίοι είναι 20 ετών και οι οποίοι νιώθουν γέροι και κάποιοι άλλοι που είναι 60 και νιώθουν νεότατοι. Λοιπόν, η δραστηριότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό το αποδεικνύει και η δράση μελών της Επιτροπής μας. Έχει μεγάλη σημασία να παραμένει κανείς δραστήριος. Στα πλαίσια της παρουσίασης της γνωμοδότησης ε, που είχε υπάρξει το 2012. Η Ευρωπαϊκή Χρονιά Αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενναίες. Θυμάμαι με τι μεγάλη ικανοποίηση είχαμε δεχθεί την πρόκληση να προχωρήσουμε στη δημιουργία σχέσεων στενότερων ανάμεσα στις νεότερες και στις παλαιότερες γενναίες και με ενδιαφέρον άκουσα τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι δεν υπήρξαν πάρα πολλά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν απέδωσε η προσπάθεια. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε στους νέους ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους και θα πρέπει να φροντίζουν τους ηλικιωμένους συγγενείς. Τα τέσσερα σημεία τα οποία προτείνατε ήταν ιδιαίτερα θετικά, ιδιαίτερα το σημείο στο οποίο επιστήσατε την προσοχή μας στη συνέχεια την οποία θα πρέπει να δώσουμε ε, στα προγράμματα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Από το 12. Αξίζει λοιπόν να υπογραμμίσουμε επίσης και τον τρόπο ελέγχου των διαρθρωτικών ταμείων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε να ενισχυθούν οι διαγενειακές σχέσεις. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη δική μας γενεά αλλά και για τις επερχόμενες. Νομίζω επίσης ότι όταν εξετάζει κανείς τις κοινωνικές επενδύσεις, λέμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ενισχυθούν και να βελτιωθούν, γιατί ε, βελτιώνουν την ζωή των ανθρώπων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες στο παρελθόν και ιδιαίτερα πριν από την κρίση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Στην Ολλανδία, σαν παράδειγμα, υπήρχαν ορισμένες επιδοτήσεις για προγόνους, οι οποίοι φρόντιζαν τα εγγόνια τους. Αυτά είναι μέσα τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε τις διαγενειακές σχέσεις, ενισχύοντας και τους ηλικιωμένους, βοηθώντας τους να παραμείνουν δραστήριοι ludziom młodych ale to co obserwuję mentorzy nie dbają o to by przygotowywać wśród ludzi młodych swoich Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους. Ludzie mądrzy, ludzie odpowiedzialni. Νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και τους νέους έτσι ώστε να γίνουν οι πραγματικοί κληρονόμοι, οι ουσιαστικοί κληρονόμοι ε, των προηγούμενων γενεών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξετάζουμε μια έκθεση που αφορά το έτος 2012, το Ευρωπαϊκό του Ενεργού Γύρανση. Το εξετάζουμε τρία χρόνια μετά και συμμερίζομαι την άποψη του προηγούμενου ομιλήτη. Φαντάζομαι ότι κάπως έχει πέσει το ενδιαφέρον. Δεύτερον, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά και θα ήθελα να μπορέσετε συζήτηση που θα έχουμε να με πείσετε για το εξής. Εάν κατάλαβα καλά τον εισηγητή, έχω την εντύπωση ότι ακόμη και παρά το γεγονό ότι λέμε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, Θέλουμε να βάλουμε τους μεγάλους ανθρώπους πάλι στην δουλειά. Το 1980, η δεκαετία του 80, που δεν είναι προϊστορία για μας, οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν στα 65 τους. Πολύ συχνά τα άτομα αυτά πέθαιναν στα επόμενα τέσσερα χρόνια και κάποιοι την ίδια χρονιά που συνταξιδοτούνταν, όπως και ο πατέρας μου. Το να ξαναβάλουμε λοιπόν όλα αυτά τα άτομα αυτής της ηλικίας πάλι στην αγορά εργασίας μου φαίνεται παράδοξο. Ανέπτυξε τέσσερα ζημία κλειδιά ο εισηγητής. Ελπίζω ότι παρανόησα. Πρώτον, θα πρέπει να κάνουμε, όπως μας είπε, τους δασκάλους κάπως, να εξυπηρετήσουμε Βγήσουμε στους πάντες ότι θα πρέπει οι μεγαλύτεροι στην ηλικία άνθρωποι να ξαναρχίσουν να δουλεύουν. Παράξενο μου φαίνεται αυτό. Δεύτερο επιχείρημα και πάλι ελπίζω ότι δεν κατάλαβα καλά μίλησε για silver economy. Δηλαδή στον κόσμο αυτό. Στην Ευρώπη αυτή που διατείνεται ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα τελικά με τους γυράσκοντες θα βγάλουμε χρήματα. Τρίτον, εφόσον μπορούμε να βγάλουμε χρήματα, θα πρέπει όλοι να υποφεληθούν. Και αυτό είναι ένα μέσο να εισαγάγουμε στην αγορά εργασίας τους νεότερους, αυτή την silver economy, δηλαδή τι κάνουμε. Τέταρτο, το κερασάκι στην τούρτα της ενιαίας σκέψης για να αποφευθεί η έκθεση αυτή να απορριφθεί, μιλούμε για διάκριση. Αλλά εδώ μιλούμε για ηλικιακή διάκριση. Ας μην βγουν από το οικονομικό μας σύστημα οι μεγαλύτεροι στην ηλικία για να μην θεωρηθούν γέροι. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε για αντίθετα επιχειρήματα να με πείσετε όταν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Αλλά πραγματικά εγώ είμαι 54 χρονών και ομολογώ ότι εκτιμώ ότι κάθε ηλικία έχει το δικαίωμα να ζει με το δικό της προνομιούχο τρόπο και όπως είπε και ο τελευταίος ομιλητής να ζει όπως θέλει για να χαίρεται. Να έχει χρόνο να κάνει χίλια πράγματα που ποτέ δεν τα κάνει όταν εργάζεται. Να αναπαύεται το δικαίωμα να ταξιδεύει. Να ανακαλύπτει τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και ίσως, όπως είπε και ένας άλλος συνάδελφος, να ασχοληθούμε σε διάφορες συλλογικές δράσεις και να βοηθήσουμε άλλα άτομα πιο μεγάλα στην ηλικία. Να ασχοληθούμε με την οικογένειά μας και κατά προτεραιότητα με τα εγγόνια μας. Φτάνουμε σε μια ηλικία στην οποία πραγματικά δικαιούμαστε να σταματήσουμε τη δουλειά μας και να σταματήσουμε να συνεισφέρουμε στην ευημερία και στον πλούτο της Ευρώπης και ο καθένας στη χώρα του βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μαγετά, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από την έκθεση αυτή εγώ, τι ε, θεωρώ σημαντικό. Αυτή η ενεργός γύρανση που αναφέρεται είναι λίγο βάρβαρη λέξη, αλλά Περί πρόκειται τελικά. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη αν ε, δούμε το προσδόκιμο ζωής για κάθε κοινωνική τάξη. Η εργατική τάξη ζει έξι χρόνια λιγότερο από τους ε, επαγγελματίε άλλων κλάδων κατά μέσον όρο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το οποίο κάνει στη ζωή του, δεν σημαίνει ότι απαραίτητο πρέπει να ξεγυρίσει στην αγορά εργασία στα 65 στα 70. Να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία, να μπορεί να ασχοληθεί με τα κοινά ώστε να δημιουργήσει και σχέσεις με άλλα άτομα. Και αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι να τονίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων γενεών. Έχουμε γονείς και παππούδες που γυράσκουν όλο και καλύτερα χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και τόσο καλύτερο και νομίζω ότι θα πρέπει να διαρωτηθούμε εμείς οι νεότεροι πώς θα τους συνοδεύσουμε με αξιοπρεπείς συνθήκες και κυρίως με την βοήθεια της ιατρικής και να δούμε πώς όλη αυτή η δομή του ιατρικού κόσμου και ό,τι τη συνοδεύει μπορεί να βοηθήσει τους ε, μεγαλύτερους να περάσουν αυτή την τελευταία φάση της ζωής τους με αξιοπρέπεια. Βεβαίω, αν λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε καλή υγεία για να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα, όχι. Αλλά όποιος επιθυμεί να σταματήσει για να ψυχαγωγείται περισσότερο και να ζει καλύτερα στο το κάνει. Αν θέλει κάποιος να έχει καλύτερη επαγγελματική ζωή. Τώρα αναφέρατε εσείς την υποψήφια των 67 ετών που είναι για την Προεδρία της Αμερικής. Χαιρετίζω τη δυναμικότητά της αν δεν αισθάνεται γριά, αλλά αν είχε ε, δουλέψει σε μια αυτοκινητοβιομηχανία για 40 χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα είχε αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική ζωή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω στον κύριο Κούκαν το λόγο τώρα για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι διότι ήδη έχουμε αρχίσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν να υιοθετηθεί η εκθεσή μου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αλλά θα κάνω απλώς κάποιες παρατηρήσεις. Με πλήσει το ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα με την ορολογία ενεργός γύρανση. Κυρίως οι Πολωνοί. Διότι εμείς και οι Πολωνοί καταλαβαίνουμε οι μεν τους δε και είναι παρεμφερείς η γλώσσα μας. Και αν μεταφράσω αυτό που είπα στα πολωνικά όλοι θα καταλάβουν τι ακριβώς εννοούμε. Τώρα, εάν ακριβώς δεν μεταφράζεται ο όρος αυτός του συνεργού γύρανσης στα πολωνικά, τι να πω. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά κρονίμια που δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε. Η εξωτερική υπηρεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μεταφραστεί ίσως, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα κρονίμι που σημαίνει αγκληματική οργάνωση. Ας μην μπούμε λοιπόν σε τέτοιου είδους θεωρήσεις. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε και η Ντανούτα. Και εγώ ξέρω πολλά άτομα τα οποία είναι 75 και είναι νέα, δυναμικά και οι αγόρια και κορίτσια που φαίνονται γέροι. Εγώ όπως λέγω η μερομηνία γέννησή σας είναι αριθμή σε ένα χαρτί. Όσον αφορά την 67 υποψήφια για την Προεδρία των ΗΠΑ, βεβαίως όλη της τη ζωή δούλεψε προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνει αυτό που θέλει να γίνει. Και κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιον ο οποίος είχε δουλέψει στην αυτοβιομηχανία με επαναληπτικές δραστηριότητες ε, επί 40 χρόνια ότι θέλει να γίνει πρόεδρος της Αμερική. 67 ε, είναι γέρος κανείς. Ο Ρίγκαν κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο με την Σοβιετική Ένωση. Πόσο χρονών ήταν ε, όταν έγινε πρόεδρος. Πάνω από 70. Άρα Μην εκφράζεστε επιτιμητικά για την κυρία αυτή. Θα εκπλαγείτε. Τώρα. Danuta's contribution, I, agree with that. Concerning Mr. Uh, Martin, I think that we shall... Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα θέματα για να καταλήξουμε. Όσον αφορά τους δύο Γάλλους συναδέλφους, η έκθεση αυτή δεν θέλει να υποχρεώσει κανέναν μεγάλη ηλικία να ξαναγυρίσει στην αγορά εργασία. Αλλά αν κάποιοι, όπως είπατε, είναι, αισθάνονται ναι και ικανοί να το κάνουν, δεν θα πρέπει να τους ε, αποθαρρύνει κανείς και να τους ε, αντικαθιστά αυτομάτως με ένα νεότερο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να μην υφίστανται διάκριση και να μην τους βάλει κανείς στο περιθώριο. Η ποιότητα της ζωής είναι σημαντική. Όντως θα πρέπει να βελτιωθεί για τα μεγαλύτερη ηλικία άτομα και ξέρουμε ότι και το παραμικρό κανείς να κάνει για αυτά τα άτομα το εκτιμούν ιδιαιτέρως και ας είμαστε πραγματικές στες. Μην ε, χαθούμε στις ε, φιλοσοφίες. Απλώς να δούμε με απλά πράγματα πώς θα βελτιωθεί η ζωή των ε, γυρασκόντων. Εάν κάποιος πιστεύει ότι ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν περισσότερο, αν θέλουν να χαρούν τη ζωή τους εκτός επαγγελματικής εργασίας, το κάνουν. Αλλά όποιος θέλει του δώσουν τη δυνατότητα και να μην ε, θεωρήσουμε ως ε, κανόνα ότι καμιά φορά στα 60 ή πολλές φορές στα 50 έτσι όπως διαμορφώνεται η τάση στη χώρα μου να τον διώχνει τον εργαζόμενο ο εργοδότης του γιατί πιστεύει ότι γέρασε. Εάν λοιπόν θέλει κάποιος να εργαστεί ας τη δώσουμε την δυνατότητα. Αν θέλει κάποιος να ψυχαγωγηθεί ή περισσότερο. Αν θέλει να συμμετάσχει σε πολιτιστικές δραστηριότητες, ας το κάνει σε κοινωνικές δραστηριότητες. Και ας τον ενθαρρύνουμε να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Είμαι σίγουρος ότι ήταν καλή η συζήτηση. Πολλά πράγματα θα διευκρινιστούν και η έκθεση θα γίνει αποκεπτή. Όχι για όλους, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά μια έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο σκέψης της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η εξέταση της έκθεσης θα γίνει στις 28 Μαΐου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 3η Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών στις 23 Ιουνίου και η υιοθέτηση ψηφοφορίας στις 15 και 16 Ιουλίου. Θα συνεχίσουμε τώρα. Στο τελευταίο θέμα στην ημερησία διάταξη, μία παρουσίαση από το Eurofund. Έκθεση για την χρήση του opt-out στην οδηγία του χρόνου εργασίας. Θα δώσω το λόγο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 Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω κάποια στοιχεία έρευνας, την οποία ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Χαίρομαι που εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Ζωής και Εργασίας uh, of the European και να σας ανεφερθώ στις χρήσεις του opt-out. Η παρουσίασή μου θα βασιστεί κυρίως στο τι έχει προηγηθεί της οδηγίας ε, χρόνου εργασίας, τις δυνατότητες εξαίρεσης από την εφαρμογή των διατάξεών της, κάποια στοιχεία της πρόσφατης έρευνας την οποία κάναμε και την οποία συνεχίζουμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την χρήση της οδηγίας opt-out, το εύρος της χρήσης του opt-out, τα επιχειρήματα που ακούγονται για το opt-out, και κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Αν δει κανεί το παρελθόν, η οδηγία του 2003, 88, η οδηγία αυτή στην ουσία θέτει τις προϋποθέσεις για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, εργασίας, στα πλαίσια της εφαρμογής των αρχών της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Οδηγία πλαίσιο 89, 39. Βασικά η οδηγία αυτή απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δώσουν εγγυήσεις για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων σχετικά με τον μέγιστο χρόνο απασχόλησης ανά εβδομάδα, τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης, και κάποια άλλα επίσης ελάχιστα επίπεδα δικαιωμάτων τα οποία καθορίζονται από την οδηγία την ίδια. Η οδηγία αυτή έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 153 της συνθήκης. Να υπογραμμίσω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ήδη τον μέγιστο χρόνο απασχόλησης, τον ανώτατο μάλλον χρόνο απασχόλησης ε, την ετήσια πληρωμένη άδεια και τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης είναι τρία στοιχεία που αποτελούν κανόνες ε, του κοινωνικού ευρωπαϊκού δικαίου. Και αναγνωρίζεται λοιπόν ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε αυτά τα τρία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω και να μην αγνοήσουμε ότι και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παρέχει την δυνατότητα για δίκαιες και σωστές συνθήκες εργασίας. Λέγει η παράγραφος 1 του άρθρου 31 ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία της του και στη παράγραφο 2 λέγει ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε ένα συγκεκριμένο ανώτατο χρονικό πλαίσιο απασχόλησης, σε καθημερινή και εβδομαδιαία ανάπαυση και σε μια πληρωμένη ε, περίοδο αδείας ανά έτος. Αυτά προβλέπει το άρθρο 31 της χάρτας. Εάν λοιπόν εμείς δούμε αυτά τα στοιχεία και πιο προσεκτικά την ίδια την οδηγία βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να εξαιρεθεί, να αποκλίνει κανείς από τις βασικές αυτές αρχές. Σύντομα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 17 αποκλήσεις για συγκεκριμένες καταστάσεις, περιπτώσεις. Το άρθρο 18, αποκλήσεις στα πλαίσια της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων. Και το άρθρο 22.1, το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα, που είναι η επιλογή των κρατών μελών να μην εφαρμόσουν το άρθρο 6, που αφορά τον μέγιστο χρόνο απασχόλησης, ο οποίος ε, λέγει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πρέπει να απασχοληθεί πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπεροριών. Εάν συγκεντρώσει κανείς την προσοχή του λοιπόν στο 31.1 ή μάλλον στο 22.1 συγγνώμη, βλέπει ότι το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη ρύθμιση εφόσον πάρει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν την σύμφωνη γνώση των εργαζομένων, ότι οι εργαζόμενοι θα συμφωνήσουν να ξεπεράσουν τις 48 ώρες, ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τους εργαζομένους αυτούς εφόσον δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν μια τέτοια ρύθμιση. Οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν καταγεγραμμένη τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να έχουν καταγραφεί και από τις επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αρχεία που δείχνουν πόσοι εργαζόμενοι επιλέγουν την απόκληση εξαίρεση σε σχέση με τον μέγιστο χρόνο απασχόλησης. το ερώτημα είναι υπάρχουν κάποια όρια σε αυτό. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο σε αυτή την δυνατότητα να εργάζεται κανείς άνω των 48 ώρων. Από ό,τι φαίνεται όχι. Η οδηγία δεν καθορίζει κάποια ανώτατα όρια εφόσον συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι για να εργαστούν άνω των 48 ώρων και δεν υπάρχει και περίοδος αναφοράς, δηλαδή σε ποια χρονική περίοδο θα υπολογιστεί κάτι τέτοιο, σε μια εβδομάδα, σε δύο μήνες, σε ένα έτος. Δεν υπάρχει διευκρίνηση ως προς αυτό για την περίοδο αναφοράς. Αν δει κανείς προσεκτικά όμως την οδηγία, μπορεί να εννοήσει ότι υπάρχουν δύο έμεσα όρια. Το πρώτο είναι 78 ώρες την εβδομάδα. γιατί ταυτόχρονα στην ίδια οδηγία οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπαύονται κατελάχιστον 90 ώρες την εβδομάδα. Αν αφαιρέσει κανείς τις 90 ώρες από τις 168 ώρες που αποτελούν τη μία εβδομάδα, δεν μπορεί να ξεπεράσει εργαζόμενος τις 78 ώρες. Και υπάρχει επίσης και ένα δεύτερο έμεσο όριο, η δυνατότητα και ο σεβασμός των αρχών της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Δηλαδή, όταν οι εθνικές αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται τα αρχεία των συμβάσεων αυτών, μπορεί να απαγορεύσουν τον εργαζόμενο να προχωρήσει σε αυτή την απασχόληση αν υπάρχουν ανησυχίες για θέματα ασφάλειας και υγείας. Και το θέμα είναι εδώ ποιες είναι αυτές οι, αυτά τα σημεία προστασίας της υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου. Δυστυχώς όμως στην πρακτική δεν είδαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σήμερα πάρα πολλές μελέτες τις οποίες διεξάγει και η ίδια Eurofound δείχνει ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα τα μεγάλα ωράρια σε μεγάλο χρονικό διάστημα και στο συχνότητα των ατυχημάτων, των λαθών, την μείωση της παραγωγικότητας, τις επαγγελματικές δυσκολίες, την πίεση και γενικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων όσο περισσότερο εργάζονται. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία λοιπόν για τις αρνητικές επιπτώσεις των ε, μακρών περιόδων απασχόλησης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το έτοιμά μας, για το έτοιμά σας συγγνώμη, να κάνουμε μια ενημέρωση, μια μελέτη επικαιροποίηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την δυνατότητα απόκλησης, το opt-out, όπως επίσης και οι εργοδότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιήσαμε ήταν ε, ε, το επίπεδο διαβούλευσης που χρησιμοποιούμε ε, συχνά με τους εθνικούς αντιπροσώπους τους οποίους έχουμε στον τομέα της, της ποιότητας στο χώρο εργασίας και της απασχόλησης θέσαμε τέσσερες ερωτήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα του opt-out. Χρησιμοποιείται η δυνατότητα αυτή. Έχετε ε, δεδομένα για τη χρήση του opt-out. Έχετε κάνει έρευνα για τις βασικές επιπτώσεις του opt-out στους εργαζομένους. Έχουν υπάρξει πρόσφατες συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Είναι μια περιορισμένη προσπάθεια αυτή την οποία κάναμε. Κάποια από τα αποτελέσματα όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτον, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις χώρες σε τρεις ομάδες. Πρώτη ομάδα είναι οι χώρες στις οποίες επιτρέπεται το opt-out και χρησιμοποιείται γενικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως τομέα και δραστηριότητας. Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά υπάρχουν 11 χώρες με επιτρεπόμενη αλλά περιορισμένη χρήση, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετωνία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία και τέλος κάποιες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Χώρες όπως η Αυστρία, η Κροατία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία. Αυτός είναι ο χάρτης λοιπόν που αντιπροσωπεύει τις τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Θα σας δώσω λίγο χρόνο για να σχηματίσετε τη δική σας εντύπωση και να δείτε τη χώρα σας. Οι περισσότερες από τις πορτοκαλί χώρες που επιτρέπουν με περιορισμένο τρόπο τις αποκλήσεις αυτές ισχύουν στον τομέα κυρίως της υγείας ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, προσωπικό στις κατεπίγουσες, στη μονάδα κατεπηγόντων κτλ. Υπάρχει επίσης ένα συσχετισμός ε, με το λεγόμενο χρόνο απασχόλησης on call, όταν πρέπει δηλαδή ο εργαζόμενος να είναι στη διάθεση της εργοδοσίας, όχι όμως το χώρο εργασίας. Κατοίκον αναμονή έτσι ώστε να κληθεί ή να είναι σε ετοιμότητα ο εργαζόμενος. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορές, αλλά ανάλογα με τη χώρα βέβαια. Θα δείτε εσείς τον κατάλογο που σας έχουμε δώσει, τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν στις διάφορες χώρες, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο χώρες, Τσεχία και Ισπανία. Οι δύο αυτές χώρες εφαρμόζουν την δυνατότητα απόκλησης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, όμως στις χώρες αυτές εφαρμόζεται μια προσωρινή νομική ρύθμιση. Αυτή η προσωρινή νομική ρύθμιση ε, έληξε χρονικά. Και τώρα λοιπόν και στην Τσεχία και στην Ισπανία δεν υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα απόκλησης. Το επόμενο ερώτημα είναι το τι γνωρίζουμε για την εκτεταμένη χρήση ε, του opt-out. Είμαστε το 2015. Οι συζητήσεις έγιναν πριν αρκετά χρόνια και δεν φαίνεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά για το εύρος της χρήσης των opt-outs, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου η μελέτη WERS, μελέτη δηλαδή των σχέσεων στο χώρο απασχόλησης το 2011 μας δίνει στοιχεία. Ακόμα και σε άλλες χώρες που είναι γενικευμένες δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Υπήρξε και μία μελέτη από την Αυστρία πρόσφατα η οποία ζητήθηκε από το ιατρικό επιμελητήριο της Αυστρίας το 2013, έκαναν 2.000 τηλεφωνικές συνεντάξεις και ζήτησαν από τους ιατρούς να μιλήσουν για τις υπερορίες τους και είδαν ότι κατά μέσο όρο σε εβδομαδία βάση ένας ιατρός δουλεύει 59 ώρες. Το 6 σε 54 το 2014. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνά προφανώς ε, την ε, ρύθμιση για την οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης. Και είπανε όλοι αυτοί οι γιατροί ότι προτιμούσαν να δουλεύουν βέβαια 42 ώρες. Ένα μεγάλο τμήμα των συμμετεχόντων, πάνω από το 60% είπαν ότι θα ήταν υπέρ μιας υποχρεωτικής μείωσης, το 76% μιας προσωρινής μείωσης επιβαλόμενης όμως. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Αυστρία που εργάζονται για πάνω από 25 ώρες συνεχώς. Λοιπόν, αυτά γνωρίζουμε προς στιγμή. Για να καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση, ελέγξαμε και την, ε, και την έρευνα για την απασχόληση το 2010 Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα opt-outs με τον αριθμό των εργαζομένων που ε, εργάζονται ε, για μεγάλες χρονικές περιόδους. Βλέπετε μπλε αριστερά τις χώρες οι οποίες έχουν γενικευμένη χρήση του μέσου απόκλησης, πορτοκαλί περιορισμένη χρήση του μέσου απόκλησης και επίσης έχετε και τον αριθμό των εργαζομένων με πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι ότι κατά μέσον όρο οι χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν το opt-out έχουν μικρό αριθμό εργαζομένων που δουλεύουν περισσότερο. Η Ρουμανία όμως και η Ελλάδα ε, πετάγονται αν θέλετε στην κορυφή. Η μακρά απασχόληση δεν είναι κάτι το οποίο συνδέεται λοιπόν με τη χρήση του opt-out, το μεγάλο ωράριο εργασίας δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την οργάνωση της αγοράς εργασίας και ακόμα και με πολιτισμικά θέματα του πόσο θεωρούνται σημαντικά τα ωράρια δηλαδή τα μεγάλα για κάποιες χώρες σε κάποιους τομείς. Στα πλαίσια τώρα των περαιτέρω συζητήσεων που γίνονται τώρα πια βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των opt-out Λίγες μόνο ή κάπως, κάποιες έχουν κάποια θέματα και η πρώτη περίπτωση είναι της Αυστρίας που έχει ενδιαφέρον διότι το Γενάρη του 2015 από 1η Ιανουαρίου δηλαδή εγκρίθηκε μια τροποποίηση του νόμου εργασίας στα νοσοκομεία που λέει δίνει την ευκαιρία δηλαδή στους γιατρούς να κάνουν opt-out, να ζητούν εξαίρεση από τις 48 ώρες αν και θέλουν μέχρι το 2020-2021 να κατέβουν από τις 60 ώρες στο όριο που περιλαμβάνει και η οδηγία, δηλαδή 48 ώρες. Είπε λοιπόν επίσημα η Αυστρία ότι δεν επιθυμεί να εφαρμόσει την ρήτρα opt-out, αλλά για πρακτικούς λόγους και επειδή υπάρχει θέμα βέβαια στον τομέα της υγείας, εφαρμόζουν τελικά το opt-out από την αρχή του χρόνου. Με πρόθεσή τους να μειώσουν το ανώτατο όριο μέχρι το 2021. Στην Κροατία πέρσι διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για μια πιο εύκαμπτη χρήση των διατάξεων του ωραρίου σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει και η περίπτωση τώρα Ιρλανδίας, Ελλάδας και Ιταλίας που παραπέμφθηκαν πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι προφανώς δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, για το ωράριο εργασίας των γιατρών στα νοσοκομεία δημόσιας υγείας, στα δημόσια δηλαδή νοσοκομεία, και έχουν μακρύτερα ωράρια. Στην Τσεχική Δημοκρατία, όπως είπα πριν, οι σχετικές ε, διατάξεις έληξαν το 2013. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι εξακολουθούν στον τομέα της υγείας να εφαρμόζονται μακρά ωράρια υγείας και πέρσι η, ε, στη Γαλλία έγινε ε, απεργία από μια κατηγορία γιατρών για λόγω υπερβολικής ε, απασχόλησης με ορισμένους να λένε ότι είχαν και πάνω από 60 ώρες την εβδομάδα. Τώρα έχω κάποιες ε, τελικές συμπερασματικές παρατηρήσεις σε σχέση με τη μελέτη. Δεν υπάρχουν πρώτα πρώτα πολλές αλλαγές από το 2010 στις χώρες που ανέφερα προηγουμένως. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει τροποποιηθεί σημαντικά. Σε ό,τι αφορά την χρήση της δυνατότητας της εξαίρεσης, πράγματι δεν γνωρίζουμε πολλά. Δεν γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε και άρα θα χρειαστεί να αναζητήσουμε και άλλες πηγές για να δούμε αν μπορούμε να αντλήσουμε από κάπου αυτές τις πληροφορίες. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να γνωρίζουμε και περισσότερα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, υπογράφονται αυτές οι ε, εξαιρέσεις συνθήκες χρόνου, πιέσους κλπ. Το άλλο που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει και μια αρνητική επίπτωση στην υγεία των εργαζόμενων στον τομέα υγείας από τα πολύ παρατεταμένα ωράρια εργασίας. Το ίδιο και ε, υπάρχουν επιπτώσεις και επί των πελατών κάθετος ασθενών. Και υπάρχουν ανάγκη, υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί εάν πραγματικά αποδίδουν τα ωράρια αυτά για τους εργοδότες ή για τα νοσοκομεία ή για τις εταιρείες. Και το άλλο που συζητούμε είναι ότι υπάρχουν πολλά ακόμα αναπάντητα ερωτήματα, ένα από τα οποία είναι και σχετικά με την κάλυψη των εξαιρεσιών αυτών. Καλύπτει μόνο τον εργαζόμενο ή καλύπτει την σύμβαση, διότι μπορεί να υπάρχουν και ε, πλήρωνες συμβάσεις εργασίας. Άρα μπορεί τελικά να καταλήξουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες διότι έχουμε εμεί εξετάσει μέχρι τότε μονάχα τις επιμέρους συμβάσεις εργασίας που έχει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι βέβαια και ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή οι της εργασίας. Έχουν πράγματι τα μέσα, έχουν τη δυνατότητα τους πόρους να ελέγξουν την εφαρμογή των εξαιρέσεων όπως είπα υπάρχει έλλειψη δεδομένων και αυτή ίσως δείχνει ότι εκεί σημειώνονται κάποια προβλήματα <clears throat> και ίσως χρειάζεται να ψάξουμε περισσότερο. Τέλος, θα είναι σημαντικό να εξετάσουμε περισσότερο και ποια είναι η αιτιολόγηση για το opt-out. Σε πολλές χώρες η συζήτηση που διεξήχθη είναι, είπαν δηλαδή, ότι αν οι άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν περισσότερο, ας δουλέψουν. Ενώ αλλού οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλέψουν παραπάνω γιατί είναι πολύ χαμηλά τα ημερομίσθια και επομένως αναγκάζονται να δουλέψουν περισσότερο για να έχουν ε, παρκές εισόδημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εν τέλει το μήνυμα πρέπει να είναι ότι πρέπει να ψάξουμε περισσότερο, άρα να κάνουμε περισσότερη έρευνα σε περισσότερο βάθος για να δούμε ποια είναι η πραγματική εφαρμογή αυτών των opt-out. Τελειώνοντας, θα δείτε στις ε, διαφάνειες επιλεγμένα, επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε σχέση με την οδηγία αλλά καθώς και, με, και σε σχέση με τα ωράρια εργασίας έχουμε και κάποια project τα οποία έρχονται την ε, έρευνα δηλαδή για τις συνθήκες εργασίας του 2015 και θα εξετάσουμε σε περισσότερο βάθος τη διασύνδεση μεταξύ των ε, παρατεταμένων ωραρίων εργασία και των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία και αλλού. Η ευχαριστώ κύριε Καμπρίτα. Αρχίζει η συζήτηση. Εντυράνκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να συζητήσει το θέμα αυτό. Απλώς θα ήθελα να κάνω κανένα δύο ερωτήσεις πραγματικά βρήκα ενδιαφέρουση. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το χάρτη που μας δείξατε, με την χρησιμοποίηση του opt-out. Είναι ενδιαφέρον το ότι είναι πάρα πολύχρωμος αυτός ο χάρτης. Κάνετε έρευνες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του opt-out σε σχέση με τα διάφορα συστήματα ε, τη, κοινωνικής ε, ασφάλισης. Επίσης, σε θέματα πολιτικής επισέρχεται πολύ αυτό το θέμα του opt-out. το έχετε συζητήσει σε διάφορες χώρες. Τι ακριβώς γίνεται. Στην ε, Ισπανία και σε άλλες χώρες κυρίως σε σχέση με το ότι κυρίως ο τομέας της ε, γεννήσει ένα τομέα στον οποίο εργάζεται περισσότερο τα διάφορα άτομα και σχέση με τη στρατηγική που ακολουθείτε, σχέση με την οδηγία αυτή για τον ωράριο εργασίας. Έχετε παρατηρήσεις ναι. όσον αφορά τι τομεακές ε, συμφωνίες. Είπατε ότι, ότι σε χώρες με περιορισμένη χρήση του opt-out υπάρχουν τομείς που εξαιρούνται έχετε σημειώσει ποιοι και με ποιο τρόπο ε, υπάρχουν εκεί τομεακές συμφωνίες. Επίσης, δεδομένου ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς ο τομέας της υγείας, έχετε κάνει καμία έρευνα για να δείτε κατά πόσον επηρεάζονται διαφορετικά από το opt-out οι άνδρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι στον τομέα αυτό, διότι ξέρουμε ότι στον τομέα της υγείας ιδιαίτερος Υπάρχουν πάρα πολλές ε, γυναίκες που εργάζονται και θα πρέπει να μου πείτε αν έχετε κάνει μια μελέτη για το πώς σε επηρεάζει αυτό ανάλογα με το φίλο τους, η κυρία Στάιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που σίγουρα έχει ε, χρησιμότητα για τις ε, συζητήσεις που θα διεξαγάγουμε. Πρώτα, αν και αυτό δεν έχει σχέση με την ενημέρωση που κάνατε, το ερώτημα κατά πόσον η ισχύουσα οδηγία και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εφαρμόζονται όντως στις χώρες μέλη. Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί πριν να ασχοληθούμε με παραπέρα ρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε, Μιλήσατε κι εσείς για τις επιπτώσεις των παρατεταμένων ωραρίων εργασίας και στους ίδιους εργαζόμενους, αλλά αν εξετάσουμε και βέβαια τον τομέα της υγείας, υπάρχουν επιπτώσεις και στους καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας. Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση για την προστασία όλων, για την αποφυγή και επαγγελματικών νόσων, αλλά βεβαίως και εφόσον πρόκειται για τη φροντίδα του ασθενούς, ενώ ο γιατρός που έχει ήδη δουλέψει 52 ώρες, ε, δύσκολα θα μπορούσα ως ασθενής να αισθάνομαι άνετα να καταλήξω στο χειρουργικό τραπέζι μπροστά του. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για άλλες ομάδε ομάδες ε, επαγγελματιών στους οποίους εμπιστευόμαστε την ίδια τη ζωή μας. Υπάρχουν όπως είπατε και εσείς πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι η χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης, του opt-out. Για μένα είναι προφανή τα οικονομικά επιχείρηματα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές. Είπατε επίσης ότι διάφορες χώρες κάνουν διαφορετική χρήση της δυνατότητας opt-out. Διαθέτεται πληροφορίες, έγγραφα, ε, πηγές για την μη συμμόρφωση με το άρθρο 22.1 που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που λένε ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να δηλώσει τη σύμφωνη ε, γνώμη του κλπ. Εν τέλει, συμφωνείτε με τη γνώμη ότι αυτή η εξαιρεση όπτα opt-out δηλαδή, με υπερβολικά παρατατωμένα ωράρια εργασίας, έρχεται σε αντίθεση και με το ίδιο το περιεχόμενο του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπασίρ. Thank you, Mr. for the work you have done on the use of opt Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε στα πλαίσια της χρήσης του opt-out στην οδηγία ε, χρόνο απασχόλησης, χρόνο εργασίας. Αυτά που είπατε δεν με εκπλήσουν εμένα και την ομάδα μου. Από την αρχή ήταν σαφές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα όπου η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι βιώσιμη ή επιθυμητή από πλευράς των κρατών μελών. Αυτό ε, φάνηκε από τον μεγάλο αριθμό των κρατών μελών που ζήτησαν το opt-out. Αυτό που επιθυμούμε σήμερα είναι ότι στις χώρες που εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία, οι μισές από τις σοβαρές, ή ε, ε, μάλλον οι μισές χώρες ε, παραβιάζουν την ίδια την νομοθεσία. Και οι χώρες όπου έχει λήξει η προσωρινή εξαίρεση δεν έχουν μπορέσει, δεν έχουν μπορέσει να εφαρμόσουν την ρύθμιση. Στην Αυστρία δεν υπάρχει opt-out, αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασία. Αν δει κανείς τα στοιχεία αυτών που εργάζονται για πάνω από 48 ώρες, θα δει ότι δεν είναι οι χώρες που χρησιμοποιούν περισσότερο την δυνατότητα του opt-out. Νομίζω ότι αυτό είναι αποκαλυπτικό. Τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξει κανείς είναι σαφή. Έχουμε έναν μεγάλο κλάδο εδώ βιομηχανιών και δραστηριοτήτων και συγκεντρώνεται θα έλεγα το φαινόμενο αυτό με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Είχαμε δυσκολίες στην υιοθέτηση και τώρα στην εφαρμογή αυτής της κακοσχεδιασμένης οδηγίας. Και αυτό αποδεικνύει ότι η λογική το ένα νούμερο κάνει για όλους δεν ισχύει. Θα συμφωνήσετε λοιπόν μαζί μου ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό ε, θα πρέπει να λαμβάνονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ γιατί συγκεντρώνετε την προσοχή σας στην επίπτωση που έχει ο χρόνος απασχόλησης στην υγεία. Υπάρχουν ορισμένοι που σκοτίστηκαν για την υγεία των εργαζομένων. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μου ζωή, στην επιχείρηση που δούλευα, υπήρχαν εργαζόμενοι που ήταν ε, πρόθυμοι να εργαστούν ακόμα περισσότερο. Θα ήταν διατεθειμένοι να εργάζονται 20-30 ώρες συνέχεια, όχι γιατί τους άρεσε, αλλά γιατί είχαν ανάγκη από χρήματα. Πρέπει να προσέχουμε, να μην χάνουμε τη ζωή μας προσπαθώντας να κερδίσουμε τα χρήματα για να ζήσουμε. Μιας και ορισμένοι κοροϊδεύουν τους εργαζομένους και τα προβλήματα υγείας, εγώ θα πάρω τους αριθμούς σας και θα μιλήσω για την επίπτωση στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Αποδεικνύεται μέσω των, ε, των γραφημάτων σας ότι οι χώρες οι οποίες ασκούν την εξαίρεση αυτή δεν είναι αυτές με την υψηλότερη παραγωγικότητα. Αποδεικνύεται δηλαδή εύκολα ότι δεν συνδέεται η παραγωγικότητα με το χρόνο απασχόλησης και το επιβεβαιώνω αυτό γιατί είμαι υπεύθυνο για μια έκθεση για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και πήγα σε οκτώ διαφορετικές χώρες, επισκέφθηκα πολλές βιομηχανίες, δεν θα με πιστέψετε, αλλά οι βιομηχανίες όπου οι εργαζόμενοι εργάζονται λιγότερο είναι και οι πιο παραγωγικές στη Βόρεια Ευρώπη. Κάποιες γερμανικές εταιρείες, κάποιες γαλλικές βιομηχανίες, κάποιες μεγάλες ισπανικές επιχειρήσεις, βελγικές επιχειρήσεις. Γιατί, γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει πολλά στο μέσο παραγωγής, στο μέσο εργασίας, χώρες που έχουν επενδύσει πολλά και στις συνθήκες εργασίας. Και ένας εργαζόμενος, τον οποίο αντιμετωπίζουμε καλά και δουλεύει κάτω από καλές συνθήκες, είναι πολύ πιο παραγωγικός. Να λοιπόν, ε, τι θα πρέπει να προσέξουμε εδώ. Συμφωνώ με αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως η Ούτα και εγώ είχα την ατυχία να αρρωστήσω, να πάω στα κατεπήγοντα σε μια χώρα που υπογραμμίσατε, στη Γαλλία. Στη Γαλλία το ιατρικό πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα οι γιατροί στα κατεπήγοντα εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Όταν φτάνετε σε μια υπηρεσία κατεπηγόντων στις 11 το βράδυ της Κυριακής Πράγματι δεν έχετε τη διάθεση να σας φροντίσει ο γιατρός, όχι γιατί είναι ανίκανος, αλλά γιατί είναι εξαντλημένος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις πληροφορίες σας. Προσοχή στην υγεία των εργαζομένων και καμία απόδειξη ότι συνδέεται η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης με το μεγάλο ωράριο εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ενημερώσω την Επιτροπή ότι η ομάδα μας οργάνωσε μια συζήτηση επί αυτού του θέματος που μας απασχολεί, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι το μέλλον της παρούσας οδηγίας. Και λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ισχύουσα οδηγία περιέχει διατάξεις οι οποίες είναι αρνητικές για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Κυρίως τι 48 εβδομαδιαίες ώρες για τέσσερις μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν εντατικά οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό η πρακτική του opt-out τελικά θα απορριθμίσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση τα ωράρια και τους ρυθμούς εργασίας. Εμείς λοιπόν ε, ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η ψυχοσωματική κίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων και ξέροντας τα αυτό να επιτρέπουμε να υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες για θέματα υγείας για τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η αρχή της συλλογική σύμβασης θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να ρυθμίζει κάποια θέματα και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα. Θα πρέπει να έχουν καλύτερη θέση οι εργαζόμενοι στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις για να προασπίζουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω το εξής. Όταν μιλούμε για ανεργία, όλο και περισσότερες προτάσεις λέγουν πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα μείωσης των ωρών ε, εργασίας αλλά διατηρώντας την ίδια αμοιβή. Και το ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, παραλλαγές και δεν γίνεται μία σωστή προσπάθεια σημαίνει ότι θα υπάρχει όλο και περισσότερη ενεργεία. Η μείωση του ωραρίου εργασίας είναι κάτι για το οποίο εδώ και χρόνια αγωνίζονται οι για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε και όχι να πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιασλόβα, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Αναλύσατε στην έρευνα που κάνατε μέχρι ποιο σημείο χρησιμοποιείται αυτή το ε, opt-out, κυρίως όταν πρόκειται για συλλογικές ε, συμβάσεις και ποια είναι τα αποτελέσματα που καταλήξατε. Ξέρετε, ήταν ο κύριος στόχος της ερευνάς σας, αλλά θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο και για τα αδύνατα σημεία, τις αδυναμίες αυτής της οδηγίας. Εκτός από το ότι ότι υπάρχουν ε, άλλα ε, σημεία που μας δημιουργούν ερωτηματικά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αφού ολοκληρώσαμε τις ερωτήσεις, να δώσω το λόγο στον κύριο Καμπρίτα για να μας δώσει σύντομες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που έχω τόσες πολλές ερωτήσεις διότι αντικατοπτρίζουν την σπουδαιότητα του θέματος το πόσο σημαντικό είναι για τις πολιτικού περιεχομένου συζητήσει. Αν αρχίσουμε με το θέμα του χάρτη, αν εξετάξουμε όλα τα ε, πρότυπα κοινωνική μερίς, όπως ελέγχθη, δεν το εξετάσαμε αυτό. Κοιτάμε ποιες είναι οι διάφορες ε, ε, σχέσεις εργαζομένων εργοδοτών από την ε, άποψη των ε, συλλογικών συμβάσεων. Και ίσως θα πρέπει αυτό να το προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά είναι καλό αυτό το οποίο μας είπατε εσείς για τα συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης και προστασίας. Ίσως όχι για την παρούσα έκθεση, αλλά το σημειώνω και είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη για να το εξετάσουμε στο μέλλον. Σε σχέση με την Ισπανία και την ε, Τσεχία και την κατάσταση που αναφέρατε, τις στρατιστικές για να μπορέσει να ε, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το ότι λύγει η προθεσμία εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Δεν έχουμε προφορήσει από την Ισπανία και εμείς θα επιμείνω για να δω αν έχουν οι συνάδελφοι κάτι την Ισπανία, αλλά για την Τσεχία ξέρουμε ότι στην πράξη ε, το opt-out στην ε, πράξη εφαρμόζεται παρά το γεγονό ότι είναι παράνομο. Από όσων ξέρουμε, ο Υπουργό Υγεία και ο Υπουργό Εργασία γνωρίζουν την κατάσταση και λαμβάνουν διάφορα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. Αλλά παρά το γεγονό ότι η νομοθεσία είναι αντίθεση, αντίθετη, το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δουλεύει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για τις διάφορες τομεακές συμφωνίες, αν αφορούν τα, θέματα, αφορούν τα θέματα αυτά και άλλους τομείς. Κυρίως ασχοληθήκαμε με τον τομέα υγείας. Οι άλλοι τομείς αφορούνται κυρίως από θέματα ε, πήγουσας ανάγκης και αν κάποιος ε, ε, ε, πρέπει να περιμένει μήπως τον καλέσουν την τελευταία στιγμή για να κάνει κάποια δουλειά. Τώρα, είναι σε κατάσταση ετοιμότητα Τώρα, ο τομέας υγείας κυρίως είναι ο τομέας τον οποίο εξετάσαμε και κυρίως όσον αφορά το πόσο επηρεάζει το θέμα αυτό τα δύο φύλλα. Προσπαθούμε να το εξετάσουμε. Σίγουρα και εδώ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και θα δούμε κατά πόσον μπορούμε το θέμα αυτό να το ε, ε συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας, πάντως ότι δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες. Τόσο αφορά την εφαρμογή. Υπάρχουν μελέτες για την ε, φορμή της ίδιας της οδηγίας. Αυτός δεν είναι δικός μας ρόλος, είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οδηγία η λέγει ότι είναι υπεύθυνη η Επιτροπή στο να, να κάνει σε, τακτά διατήματα αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία αυτή όσον αφορά το ωράριο εργασία. Και ξέρω ότι για την εφαρμογή αυτού του θέματο έγιναν δύο μεγάλε μελέτε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματά του όταν ολοκληρωθούν οι επιπτώσεις στην ε, τομέα της υγείας με το opt-out. Η ερώτηση που αξίζει χιλιά δολάρια. Δηλαδή, κατά πόσον θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, την οποία 11 ή 12 χώρες επιτρέπουν στο σύστημα υγεία τους το ιατρικό και παραϊατρικό ε, προσωπικό να εργάζονται πέραν των ε, προβλεπομένων εβδομαδιαίων ωρών. Αυτό είναι κάτι που αφορά επίσης και τα θέματα κοινής ε, των εργαζομένων. Και μην ξεχνούμε ότι οι γιατροί δεν έχουν πελάτες, έχουν ασθενείς. Θα ήθελα να την προσοχή σας στο γεγονό ότι σε κάποιες χώρες ξέρουμε ότι οι νέοι γιατροί στην αρχή της σταδιοδρομίας τους θέλουν να δουλεύουν περισσότερο για να μπορέσουν να αποκτήσουν πείρα το συντομότερο δυνατό και για να αυξηθεί η αμοιβή τους. Θέλει λοιπόν ένα νέος γιατρός να εργαστεί περισσότερο. Ποιο μπορεί να τον προστατεύσει λοιπόν από τον ε, εαυτό τους αν δουλεύουν πάρα πολλέ ώρες. Δεδομένου ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ατομικό opt-out. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ε, απευθείας να παίξουν ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, μου ζητήσατε στοιχεία για το αν κάποιος ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν σε θέματα opt-out. Δεν έχω, δεν έχω τέτοιου ισχύει Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Κομισιόν είναι Θα πρέπει να δούμε κατά πώς πρώτα απ' όλα γίνεται και οι εθνικές ε, διατάξεις στην κάθε εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του ε, συστήματος αυτό στην πράξη είναι πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία και πώς το opt-out. Μπορώ να σας δώσω κανένα δυο παραδείγματα. Ε, εάν κάποιος θέλει να βελτιώσει τη σταδιοδρομία του, καμιά φορά υφίσταται πιέσεις και θέλει και ο ίδιος να εργαστεί περισσότερο για να φανεί ότι εργάζεται σκληρά και να πάρει προαγωγή. Μπορεί εδώ να υπάρχει το οικονομικό κριτήριο, αλλά όχι απολύτως, δεδομένου ότι την χάνει και μεγαλύτερης αναγνώρισης όταν πάρει προαγωγή και γίνει κάποιος. Τώρα, παραβίαση του χαρτί. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ. Να απαντήσω. Ουδέν σχόλιο, λοιπόν, περί αυτού. Κοινοτική νομοθεσία αν δεν θα πρέπει η νομοθεσία να είναι νομοθεσία κάθε κράτους μέλους χωριστά. Τι λέγεται τώρα σύμφωνα με την οδηγία. Ο κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αν θέλει να εφαρμόσει αυτό ή όχι. Αποφασίζει η ίδια. Και για τις προθέσεις τους τα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πώς γίνεται η εφαρμογή της οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος, πρέπει να δούμε εάν στην πράξη ακολουθούνται οι διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία. Σχέση με την ανταγωνιστικότητα, εξαιρετική ερώτηση. Εμείς όμως ειλικρινά ασχολούμεθα με το περιεχόμενο της οδηγίας, η οργάνωση του χρόνου εργασίας, θέματα υγείας και ασφάλειας. Η ανταγωνιστικότητα είναι άλλο θέμα. Αλλά ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ε, άλλης μελέτης. Οι επιπτώσεις των πολλών ωρών εργασίας και η ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς αναφέρατε κάποιο παράδειγμα από την βιομηχανία. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες συλλογικέ ε, συμβάσεις που προβλέπουν 35 ώρες εβδομαδιαία εργασία. Αν θέλει κανείς να γίνει ανταγωνιστικός, να κάνει κάτι άλλο, υπησέρχονται και άλλα θέματα. Οι ιατροί στην Γαλλία είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ίσως όμως όχι μόνο και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Τσεχία. Είναι σαφές λοιπόν ότι σε πάρα πολλές χώρες τίθεται το θέμα των ιατρών που εργάζονται πάρα πάρα πολλές ώρες. Και τέλος, δεν θα ήθελα να αποφύγω κάποιες ερωτήσεις. Ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων που έθεσε ένας συνάδελφός σας είναι κάτι το οποίο δεν αγνοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτονται από το άρθρο 18 της οδηγίας. Το άρθρο 18 λέγει ότι μέσω των συλλογικών συμβάσεων οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να αποφασίσουν να αποκλίνουν από αυτά τα οποία λέει η εβδομάδα, αλλά όχι από τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης. Έτσι λοιπόν όταν ερχόμαστε στα υπόλοιπα θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσουν θετικά ε, σε σχέση όμως με τις ατομικές επιλογές ε, νομίζω ότι ε, δυστυχώς δεν χρειάζεται παρά ένα μικρό χαρτί και με μια ατομική συμφωνία ο εργαζόμενος λέγει ότι θα μπορέσει να εργαστεί άνω των 48 ώρων. Τώρα αν δεν κάνω λάθος γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα ισχυρός στα νομικά όταν υπάρχουν ατομικές ρυθμίσεις και τομιακές ρυθμίσεις ή και επιχειρησιακές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ότι θα εργάζονται περισσότερο οι εργαζόμενοι, τότε οι κοινωνικοί εταίροι στην ουσία αποκλείονται, για να σας το πω απλά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πήραμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τις οποίες είχαμε θέσει. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να προσθέσει. Όχι από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεν θέλει. Σας ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα φορτισμένο πολιτικά και με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε αυτά τα οποία μας είπε ο ερευνητής της Eurofound και τα στοιχεία της Eurofound. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσε η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 7 Μαΐου εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση.